Absolutely, absolutely. It, it does take uh, usually. Okay. Here we go. Λοιπόν, άντε, ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, καθίστε. Το πρόβλημα των μικροφώνων, από ό,τι φαίνεται, λύθηκε, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ που ήρθατε. Να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται στο διαδίκτυο και για τη διερμηνία προτεραιότητα δίνεται στα τακτικά μέλη και στις γλώσσες τους. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την έγκριση των πρακτικών της 19ης ε, Μαρτίου και να σας παρακαλέσω αν έχετε παρατηρήσεις ε, για τα πρακτικά μέχρι το τέλος της ε, συνεδρίασης. Και το περνάμε στην σημερινή και αυριανή ημερήσια διάταξη. Σήμερα και αύριο. Ναι, αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, έγκρινε τη μερίσια διάταξη. Και θα ήθελα να περάσουμε κατευθείαν στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης το μέλλον του ελέγχου συμβατικών όπλων στην Ευρώπη και με χαρά σας παρουσιάζω δύο διακεκριμένους πανελίστες. Πρώτα τον κύριο Ρόμπιν Μόσινκοφ, που είναι επικεφαλής ε, του σχετικού τμήματος των ΟΑΣΕ. Και τον κύριο Βίλιαμ Άλμπερκ που εκπροσωπεί το ανάλογο τμήμα του ΝΑΤΟ, επίσης που αφορά τον έλεγχο συμβατικών όπλων. Πολύ επίκαιρα θέματα σήμερα. Μιλάμε λοιπόν για το μέλλον και θα ακούσουμε άρα την τρέχουσα κατάσταση ελέγχου συμβατικών όπλων και άρα σενάρια τα οποία θα ήθελα να παρουσιάσουν οι προσκεκλημένοι μας χωρίς ε, περαιτέρω χρόνο τριβή να δώσω τον λόγο στον κύριο Μοσίνκοφ και μετά στον κύριο Άλμπερκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε που ε, έχουμε και εμείς την τιμή να είμαστε εδώ και να μιλήσουμε για τον έλεγχο όπλων. Το να μιλήσουμε για το μέλλον του ελέγχου όπλων είναι βεβαίω μια υπερβολή. Δύσκολα μπορεί κανείς να προβλέψει το μέλλον. Ε, καλό είναι να κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή. Μια από έλεγχος όπλων έχει μια μεγάλη ιστορία στην Ευρώπη και καλό είναι να... Θα κάνουμε και κάποιες προβολές βεβαίως, αλλά θα ήθελα να αφαιρθώ στο τι κάνει ο ΟΣΕ. Λοιπόν, κοιτώντας το πώς ε, λειτουργεί ο ΑΣΕ και τις διάφορες διαστάσεις της ε, συνολικής ε, προσέγγισης, προφανώς Υπάρχουν τρεις ε, διαφορετικές διαστάσεις, η πολιτικο-στρατιωτική, η οικονομική και περιβαλλοντική και η ανθρώπινη διάσταση. Η πρώτη διάσταση βεβαίως διαχωρίστηκε ε, πριν από χρόνια στο στρατιωτικό και στο πολιτικό σκέλος. Έχουμε βεβαίως και το θέμα της αντιτρομοκρατίας, ε, κυβερνοασφάλειες, αστυνομικά ζητήματα, ασφάλεια συνόρων, ναρκωτικά σε αυτό επικεντρώνεται το μη στρατιωτικό σκέλος. Ε, μιλώντας όμως σήμερα για τον έλεγχο όπλων, αν δούμε τα πράγματα ιστορικά, αυτά ξεκίνησαν ε, ε, η τελική πράξη του Ελσίνκη δηλαδή το 1975 δεν προέκυψε ξαφνικά ή σε λίγου μήνε, ήταν κάτι το μακροχρόνιο που χρειάστηκε πολλά χρόνια, είχε ξεκινήσει το 1969 και είχε προταθεί από τη Σοβιετική Ένωση ε, να υπάρξει δηλαδή μια διάσκεψη για την ασφάλεια στην Ευρώπη και καλό να το σκεφτούμε γιατί τελικά χρειάστηκαν ε, έξι χρόνια και υπήρχε ο δεκάλογος ε, του Ελσίνκη ε, που ανέφερε ακριβώς κάποιες αξίες ε, με βάση τις τότε απειλές μεταξύ των δύο μπλοκ που επηρέαζαν προφανώς ε, και το ΝΑΤΟ με κυρίαρχες της ΙΠΑ και την Σοβιετική Ένωση και έτσι ξεκίνησαν αυτές οι αξίες οι οποίες θα έλεγα ότι υπάρχουν 20-30 χρόνια μετά. Η πρώτη λοιπόν αυτή τελική πράξη επικεντρώθηκε στον έλεγχο όπλων, τα πολιτικά και στρατιωτικά σκέλη και αυτές οι πτυχές της ασφάλειας και οι αρχές ε, βεβαίως ε, που καθοδηγούσαν τα κράτη βασίζονταν στην εμπιστοσύνη αλλά έπρεπε να υπάρξουν κάποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ε, το πρώτο λοιπόν ήταν να υπάρχει μια ανταλλαγή πληροφοριών. Το τι έχει δηλαδή ο καθένας ε, ως οπλισμό που απειλεί την άλλη πλευρά. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Ειδικά τη δεκαετία του 80 και 90 έγιναν κάποιες ρυθμίσεις που ισχύουν και σήμερα. Εδώ πέρα έχουμε τα τρία ακρονίμια που θα χρησιμοποιήσω. Το πρώτο είναι οι συμβατικές δυνάμεις ε, στην Ευρώπη, η σύνθηκη CFE, η συνθήκη ανοιχτών ουρανών και το έγγραφο της Βιέννης. Το πρώτα δύο είναι πραγματικές συνθήκες που κυρώθηκαν και είναι νομικά δεσμευτικές. Το έγγραφο της Βιέννης είναι πολιτικά δεσμευτικό. Και επίσης ε, στην εισαγωγή ε, είπατε ότι θα μιλήσουμε στην, ε, για τη συνθήκη CFE η συνθήκη CFE ανεστάλλει από ένα κράτος μέλος. Ο ΑΣΕ δεν είναι οργανισμός, ε, ε, γι' αυτό έχουμε συμμετέχοντα μέλη, όχι κράτη-μέλη, αλλά τα μέλη τα οποία κύρωσαν την συνθήκη για τις σημαντικές δυνάμεις στην Ευρώπη, 30, ε, σας κοιτάω για τον αριθμό. Γιατί μπερδεύω τους ανοιχτούς ουρανούς με την CFE. 30 και 34. Λοιπόν, οι 30 χώρες που συνυπέγραψαν την ε, συνθήκη ΣΥΕΦΗ ε, τελικά έγιναν 29 το 2007. Έχουμε λοιπόν 29 χώρες. Ε, αν αναρωτιέστε, η Ρωσία ανέστηλε την συνθήκη και άλλες χώρες ακολούθησαν το 2011 όταν δεν υπήρχε αντίδραση για να υπάρχει αμοιβαιότητα, δηλαδή δεν αντέλασαν συμφωνίες με τη Ρωσία. Οπότε η συνθήκη αυτή βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Η συνθήκη για τους ανοιχτούς ουρανούς ε, λειτουργεί αρκετά καλά από την άλλη. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το πώς μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί στην τρέχουσα πραγματικότητα, δουλεύοντας με διάφορους αισθητήρε, αλλά αφορά ολόκληρη την επικράτεια ε, των ε, λοιπόν της για υπερπτήσει. Οπότε και αυτό είναι ένα μέτρο εμπιστοσύνη και μπορεί κανεί να επαληθεύσει το τι γίνεται και η συνθήκη για τους ανοιχτούς ε, βοηθάει να διακρίνουμε την αλήθεια. Αν δούμε λοιπόν τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη ε, που επινοήθηκαν μέσω του εγγράφου της Βιέννης ε, στη δεκαετία του 90 μέσω του εγγράφου Μαδρίτης και Στοχόλμης, τώρα λέγεται εγγραφό της Βιέννης. Το 1999 είχαμε την πρώτη του εκδοχή και αφορούσε ακριβώς τις δυνατότητες, όχι τόσο δηλαδή τις μειώσεις ε, των όπλων, μείωνε τα όπλα σε μεγάλο βαθμό, ε, τα θωρακισμένα στοιχεία πυροβολικού, μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Όχι τόσο πολύ όμως το έγγραφο της Βιέννης, το οποίο είχε στόχο το δυναμικό κομμάτι, δηλαδή ασκήσεις επιχειρήσεις που προκαλούσαν ανησυχίε. στο έγγραφο της Βιέννης δηλαδή δίνει ευκαιρίες να πάει κανείς σε μια άλλη χώρα και να κάνει μια επιθεώρηση ή αξιολόγηση όπως τη λέμε, ε, περιορισμένη μεν. Ε, μιλάμε για τρεις ε, ποσοστώσεις ανά έτος, ανά χώρα. Οπότε έχει τα ωριά της, αλλά δίνει την δυνατότητα σε όλα τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίε για τον σχεδιασμό, τις αμυντικές δαπάνες και είναι μια ένδειξη για το τι συμβαίνει στο μέλλον. Οπότε αν δείτε το μέλλον, το που ξοδεύουν τα λεφτά, νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντικό το έγγραφο της Βιέννης. Το έγγραφο της Βιέννης παρακολουθείτε στενά από το Φόρουμ για την ε, Συνεργασία της Ασφάλειας, το δικό μου το τμήμα, το οποίο συνέρχεται κάθε εβδομάδα και μιλάει για την εφαρμογή μεταξύ άλλων αυτού του εγγράφου της Βιέννης. Έχει μια ευρεία εντολή, ε, εργάζεται και επί νέων συμφωνιών, οι αλλαγών συμφιστάμενες συμφωνίες και τα 57 κράτη που συμμετέχουν ε, συναντώνται. Η Προεδρία αλλάζει τρεις φορές το χρόνο, και θα έχουμε ρωσική προεδρία τους επόμενους τέσσερις μήνες. στο πρόγραμμα συζητάμε επίκαιρα ζητήματα που μπορεί να αφορούν είτε την μη διάδοση είτε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για όπλα μαζικής καταστροφής. Ε, είναι συνεχής οι, εβδομάδες, οι συζητήσεις κάθε εβδομάδα και υπάρχει ακριβώς ε, μια όθηση για να αλλάξει η στασιμότητα στα ευρωπαϊκά ζητήματα ασφαλείας. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά έγγραφα που απασχολούν το φόρουμ μας. Ε, δεν θα τα αναφέρω όλα, αλλά έχετε μία εικόνα για το τι μέτρα έχουμε που περιλαμβάνουν ανταλλαγέ πληροφοριών, συζητήσεις, το πώς γίνεται η εφαρμογή και το εάν απαιτούνται ανταλλαγέ. Τώρα, το βάρος το οποίο ε, δεκαετία του 1990 αφορούσε τον έλεγχο όπλων και τη μείωση όπλων στην Ευρώπη ε, έχει επιτύχει τον στόχο της. Ε, δηλαδή, οι βασικοί προμηθευτές όπλων είναι πολύ κάτω από τα επίπεδα που είχαμε συμφωνήσει τότε και ο έλεγχος όπλων με την κλασική έννοια, δηλαδή της μείωσης ε, του οπλισμού και ενό συγκεκριμένου επίπεδου το οποίο έρχεται για την άμυνα, ε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι το έχουμε επιτύχει. Προφανώς αυτό δεν ισχύει με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που θα έπρεπε να έχουν τα κράτη-μέλη ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά την τελευταία δέκα ετία το βάρος έχει πέσει από τα βαρέα όπλα περισσότερο στο τι έχουν τα κράτη ε, ως συγκρούσεις ε, μεταξύ τους και τις απειλές από μη κρατικούς δρόντες. Και έτσι περνάμε σε ένα μηχανισμό για την μείωση των ελαφρών όπλων ε, και των μικρών όπλων και των πυρομαχικών. Θα έλεγα πως η μισή μου ημέρα αφιερώνεται σε αυτό, δηλαδή στο πώς θα μειώσουμε τον όγκο των μικρών όπλων και πυρομαχικών. Ξέρω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει πολλά και στο άμεσο περιβάλλον της για να μειώσει την απειλή και της παράνομης διακίνησης και του μη ελέγχου των μικρών όπλων. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν σχετίζεται για κάποιους άμεσα με τον έλεγχο συμβατικών όπλων, αλλά είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όταν οι άλλες πτυχές απέχουν ακόμα από συμφωνία. Και έρχομαι σχεδόν στην τελευταία διαφάνεια, η οποία αφορά τις προκλήσεις που έχουμε με τον έλεγχο συμβατικών όπλων. Ανέφερα ήδη το ότι η Ρωσία αποχώρησε από τη συνθήκη ΣΥΕΦΗ, e, που σημαίνει ότι δεν μπορούν τα μέρη να εξετάσουν το ένα το άλλο, γιατί βεβαίως η συνθήκη είχε στόχο την καταμέτρηση των όπλων, σας είπα τεθωρακισμένα, στοιχεία πυροβολικό κτλ. Ο εξυγχρονισμός ε, του εγγράφου της Βιέννης για να λάβει υπόψη και τις συγχρονές δυνατότητες και τα μαθήματα των τελευταίων 10-20 ετών για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί περισσότερη εμπιστοσύνη εξετώνοντας τις ενόπλες δυνάμεις. Έχουμε τις συζητήσεις για τους ανοιχτούς ουρανούς για το πώς θα εξυγχρονιστούν οι αισθητήρε ε, να γίνουν ψηφιακοί, κάτι το οποίο ανησυχεί πολλά κρατημέλη. Προφανώς το θέμα της Ουκρανίας έχει σημαδέψει τις συζητήσεις στην Βιέννη για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον έλεγχο όπλων. Η αντίληψη απειλών και το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές ε, διαφέρουν πάρα πολύ και δεν είναι εύκολο να καταλήξουμε σε μία άποψη για το τι μορφή θα έχουν αυτά. Υπάρχουν επίσης πολλές ε, συγκρούσεις που υπάρχουν εδώ και καιρό στον Κάφκασο, στη Μολδαβία, στη Γεωργία που δεν έχουν επιληθεί επί σειρά ετών και δεν είναι εύκολο να προχωρήσουμε όταν έχουμε αυτή την κατάσταση. Προφανώς οι σχέσεις ΙΠΑ και Ρωσίας επηρεάζουν πολύ το πώς βλέπουμε το θέμα του ελέγχου όπλων, αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι Υπάρχει υπουργική διάσκεψη υπουργών εξωτερικών κάθε χρόνο. Πέρσι έγινε στο Αμβούργο και υπήρχε μια συμφωνία τουλάχιστον να γίνει ένας διάλογος ελεγχού όπλων ή για μια αρχιτεκτονική ασφαλεία της, ασφαλείας της Ένωσης στα γνωστά φόρα όπως το δικό μας ε, είχαμε λοιπόν ε, την πρώτη συνάντηση σε επίπεδο πρωτευουσών την προηγούμενη Παρασκευή, είχαμε διάφορες απόψεις, αλλά τουλάχιστον ξεκίνησε μια διαδικασία για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συμβάσουμε τις διαφορετικές αντιλήψεις περί απειλής και να πάμε σε συζητήσεις στρατιωτικού δόγματος, το πώς είναι τοποθετημένες οι δυνάμεις και το τι μπορούμε να κάνουμε και με την συνθήκη CFE που έχει τελματώσει και με άλλες συμφωνίες όπως το έγγραφο της Βιέννης το οποίο είναι πολιτικά δεσμευτικό όπως είπα και ίσως είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί εκεί η πρόοδος. Εν ολίγης, αυτά ήθελα να σας πω ως εισαγωγή. Αυτή τη δουλειά κάνουμε και ευχαριστώ να δεχτώ ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα σας προτείνω τώρα να έχουμε τις ερωταπαντήσεις. Μετά. Αλλά πρώτα πρώτα να λάβει το λόγο ο κύριος Άλμπεργκ, αν θέλει. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να μιλήσω για αυτό το θέμα. Είναι, πολύ, είναι ένα θέμα το οποίο δεν το ξέρουν πολύ. Γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσω να κάνω ένα μικρό ιστορικό πριν μπούμε στη σημερινή κατάσταση. Ε, όμως ε, ο έλεγχος όπλων ε, δεν είναι γνωστός, ή το ιστορικό αυτού δεν είναι γνωστό σε πολλούς. Εγώ είμαι στον ΝΑΤΟ εδώ και τα 4,5 χρόνια και εξετάσουμε το παρελθόν ε, μέσα από τα, το οπτικό πρίσμα του παρόντος. Η κατάσταση ήταν ασταθής, υπήρχαν πολλοί παράμετροι, πολλές παράμετροι και υπήρχε περίπτωση ε, όλος ο κόσμος να περάσει και να ζήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλοι θυμόνταν ε, τι φρίκες των πολέμων ε, και το ενδεχόμενο της, του αφανισμού της ανθρωπότητας. Μία σειρά από κρίσεις, τις δύο κρίσεις του Βερολίνου, του, τον κόσμο, στην Τσεχοσλοβακία, Μέση Ανατολή, Κούβα κτλ. έμοιαζε ότι ο κόσμος θα αφανιστεί σύντομα. Το 1967 ο Βέλγος ε, Υπουργό ε, Εξωτερικών, ο Πιουρ Χαλμέλ, μετά έγινε και Πρωθυπουργό, αποφάσισε να ε, ξαναθέσει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Γιατί είχε δημιουργηθεί το, το ΝΑΤΟ. Ε, ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να υπερασπίζεται τα μέλη του, είπαν λοιπόν, ε, ούτω ώστε να αισθάνονται ασφαλή. Και με βάση αυτή την αίσθηση ασφάλεια να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν την Σοβιετική Ένωση, ούτω ώστε να λύσουν τι πολιτικέ κρίσει για να εξασφαλιστεί η ειρήνη στο μεταξύ να χρησιμοποιήσουν τον έλεγχο των όπλων, τον αφοπλισμό και το μη πολλαπλασιασμό, ούτως ώστε να υπάρξει ειρήνη και ασφάλεια ε, με τις λιγότερες δυνατές δυνάμεις. Δεν, θέλουν, δεν θέλει κανένας ε, αγώνα για τα όπλα. Και τη δεκαετία του 60 αυτός ο αγώνας για να αποκτήσει ο καθένας ε, περισσότερα όπλα έγινε όλο και... Ο ανταγωνισμό των εξοπλισμών ήταν όλο και πιο ακριβώς. Προσπαθούσαμε λοιπόν με το διάλογο να σταματήσουμε τον ψυχρό πόλεμο. Από αυτή την απόφαση ε, προέκυψαν τρει άξονε δουλειά. Καταρχά, όπω είπε ο Ρόμπιν, να δεχτούμε την Σοβιετική προσφορά για ειρηνευτικέ ε, συνομιλίε. Και έτσι δημιουργήθηκε η ε, ΟΑΣΑ και το Φόρουμ της Βιέννας και προσπαθήσαμε Κανένα να μην έχει το πλεονέκτημα σε δυνάμει, ούτω ώστε ε, να μην κάνει επιθέσει εθνικιαστικέ κτλ. Ε, Επίση, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ ήθελαν να ξέρουν ότι οι ΗΠΑ δεν θα πουλούσαν ξαφνικά ε, την Ευρώπη στους Σοβιετικούς, σε μυστικέ συμφωνίε. Μερικέ φορέ φάνηκε ότι θα γίνει αυτό, ειδικά κατά τι διαπραγματεύσει του ΣΟΛΤ ε, στις αρχές δεκαετία του 1970. Επομένως, οι σύμμαχοι ήθελαν να μπορούν να μιλάνε και αυτοί για τις διμερείς συμφωνίες Αμερικανών Σοβιετικών. Λοιπόν, πώς ανεπλάκει το ΝΑΤΟ τώρα. Ε, οι πρέσβοι στο ΝΑΤΟ ε, συζητούσαν κάθε ε, βασικό σχέδιο συμφωνίας. Παραδείγματο χάρη σύμβαση για τα φιλολογικά όπλα, συμβατικά όπλα κτλ. Όλα περνούσαν από το αρχηγείο του ΝΑΤΟ και σταματούσαν ε, στη Γενέβη τις συνομιλίες για να εξετάσουν ε, λιγάκι αυτές τις συμφωνίες. Επίσης στο ΝΑΤΟ υπάρχει μια ειδική ε, επιτροπή για να συζητά τις διμερείς συμφωνίες Σοβιετικής Ένωσης, ΗΠΑ, η συμβουλευτική αυτή ομάδα όπως λεγόταν. Επίσης είχαμε μια ε, ομάδα υψηλού επίπεδου που εξακολουθεί να υπάρχει και υπήρχε και υπάρχει σήμερα, εξακολουθεί να υπάρχει για τα συμβατικά όπλα και μια ομάδα πυρηνικού σχεδιασμού που ο κόσμος θεωρεί ότι αυτή συνεισέφερε στον αφοπλισμό. Αλλά τη χρονιά μετά την... Ε, σταμάτησε κάποια χρονιά, ας πούμε, ε, το 1967, από εκεί και πέρα να μειώνεται ο αριθμός των όπλων. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλήσει με του ε, συμμάχου, ε, αφού μίλησαν οι Αμερικανοί, αποφάσισαν ότι χρειάζονται τόσα πολλά όπλα για να υπερασπιστούν, τους, για να υπερασπιστούν οποιαδήποτε στιγμή, πούμε, του συμμάχου. Επομένω, ε, τι κάνανε λοιπόν με τον έλεγχο των όπλων. Ε, όταν οι Αμερικάνοι και οι Σοβιετικοί είχαν κοινό συμφέρον να αποφύγουν τον ε, κατατύχη πόλεμο, τότε αυτό ο έλεγχο των όπλων λειτουργεί καλά και όλοι προσπαθούσαν να, ενώ όταν όλοι προσπαθούσαν να κάνουν το δικό του, α πούμε, τίποτα δεν πάει καλά. Ε, είχαμε λοιπόν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ε, εδώ ε, υπάρχει η έννοια της, του στρατιωτικά σημαντικό. Θα πρέπει να είναι δεσμευτικό για όλα τα μέρη, να υπάρχει αμοιβαιότητα και να υπάρχει επαλήθευση. Δηλαδή όλοι να κάνουν αυτό που λένε θα κάνουν. με αυτόν τον τρόπο ε, μπορεί να ανοιχνεύσει σημάδια πιθανή ε, ένοπλη σύραξη και μη συμμόρφωση. Επίση, είχαμε και το φόρουμ, την ΟΑΣΕ, ε, όπου ελέγχαμε και είπαμε ότι και εκεί ελέγχαμε, ας πούμε, ότι ο καθένας δεν κάνει κάτι το οποίο θα μπορέσει να οδηγήσει σε πόλεμο. Όμως, ο έλεγχος αυτός ε, των όπλων δεν είναι κάτι το μαγικό, ας πούμε. Απλώς σου δίνει κάποιο χρόνο προειδοποίησης. Και επίσης θα πρέπει να λειτουργεί παράλληλα με τις, υπηρεσί... με τις μυστικές υπηρεσίες. Θα πρέπει ε, να εμπλακούν και εκεί οι στρατιωτικοί. Ένα άλλο πράγμα που κάνει ε, η ΟΑΣΕ είναι αυτό. Ε, η συνθήκη του, του 1970 ήταν ένα βήμα προς τα πίσω, ένα βήμα ας πούμε χαλάρωσης. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση. Τα καλά νέα είναι η συμφωνία για το Ιράν, θαυμάσια συμφωνία, ε, ούτως ώστε να υπάρχει επαλήθευση για οτιδήποτε γίνεται, συνεργασία για, την, ε, για το μη πολλαπλασιασμό, και η φάση της ε, εφαρμογής του ΣΤΑΤ. Το κακό όμως ποιο είναι. Ότι ο έλεγχος των όπλων στην ευρωατλαντική περιοχή είναι υπό απειλή. Το INF, ε, οι Ρώσοι δεν εφαρμόζουν, τα άλλα 29 μέρη εφαρμόζουν τα μεταξύ του συμφωνηθέντα. Γεωργία, Αζαρμπαϊτζάν, η συμμαχή του ΝΑΤΟ, Ουκρανία, Λευκορωσία, όλοι θα πρέπει να καλύπτονται από την ε, συνθήκη περιορισμού, ακόμα και αν η Ρωσία δεν συμφωνεί. Και επίση και το παγκόσμιο καθεστώ NPT ε, είναι που απειλεί του μη πολλαπλασιασμού, δηλαδή των ε, όπλων. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Τι γίνεται στη Νέα Υόρκη τώρα. Έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος, ε, θα ανοίξει ο δεύτερος. Φυσικά έχουμε την Ινδία, το Πακιστάν, τη Βόρεια Κορέα. Όλα αυτά είναι υπό απειλή την ε, συμφωνία του Βουκουρεστίου, επίση που απειλεί, τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Μπορούμε να επανέλθουμε στα βασικά, ε, να αισθάνονται πιο ασφαλείς οι, οι σύμμαχοι και να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε διάλογο με τη Ρωσία. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι μονίμως προσπαθούμε να συνδιαλεγόμαστε με τη Ρωσία. Το τέλη Μαρτίου κάναμε ε, μία συνάντηση, ο στρατηγός Ουρλόφ ε, μίλησαν για τις, και άλλοι Ρώσοι, είπαν τις απόψεις τους για τα θέματα αυτά της, ε, της ανάπτυξης ε, στρατιωτικού δυναμικού κτλ. Συμμετείχαν και τα υπόλοιπα κράτη. Ο διαρθωμένος διάλογος τώρα. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα. Ο συνάδελφος σας ανέφερε γι' αυτό, αλλά να σας πω ότι είναι πραγματική ευκαιρία για τον έλεγχο των συμβατικών όπλων στην Ευρώπη ο Γερμανός Υπουργός Μάιρ έκανε πρόταση στην εφημερίδα ότι θα πρέπει να υπάρχει διάλογος με τη Ρωσία και θα μπορούσαμε μετά το διάλογο αυτό να επιτύχουμε πρόοδο στον έλεγχο των όπλων. Ε, το Δεκέμβριο στην Υπουργική του και οι 57 χώρε ε, συμφώνησαν να ξεκινήσουν το διαρθωμένο διάλογο με βάση αυτή την πρόταση, ούτω ώστε να δούμε τι θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Ε, δημιούργησαν μια ομάδα ανοιχτή. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά, όπω είπε και ο Ρόμπερτ, την Παρασκευή 7 Απριλίου και η συνάντηση ήταν αρκετή επιτυχία. Ε, Κανένα δεν έφυγε κραυγάζοντα έξω από το δωμάτιο. Ξε, ξεπέρασαν τα, τα, τα κλασικά του διαλόγου, ας πούμε. Υπάρχουν δυνατότητε αν έρθει η Ρωσία και μιλήσει. Αν έρθει τραπέζι. Τώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι θα γίνει. 4 και 5 Μαΐου θα γίνει μια συνάντηση για το στρατιωτικό δόγμα ε, στρατιωτικοί ε, υπό την Αυστριακή Προεδρία θα συζητήσουν για να συζητήσουν για το στρατιωτικό δόγμα. Και κάθε μία από τι συμμετέχουσε χώρε θα μπορεί να μιλήσει για τι δυνάμει, της, ε, τα σχέδιά τη, γιατί οι δυνάμεις τη κινούνται με τον τρόπο που κινούνται, ποιο είναι το μέλλον αυτής τη ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων κτλ. Και αν κατά πόσο συνάδει με τους στόχους κτλ. Και του τους στόχου. στόχους. Και ε, τι 6 Ιουνίου θα περάσουμε στον ενισχυμένο διάλογο για την ε, πραγματική ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων αυτή καθεαυτή. Στις 11 Ιουλίου μετά θα γίνει ε, η άτυπη υπουργική του ΑΣΕ για να δούμε πού έχουμε φτάσει, ε, ποιος εποπτεύει αυτή την διαδικασία. Είναι ένας πρέσβης ε, από τη Γερμανία, ο οποίος θα κάνει και συστάσει για τα επόμενα βήματα. Αλλά πάνω απ' όλα δεν μπορούμε να κάνουμε συμβασμού πάνω σε ένα παγκόσμιο σύστημα που να βασίζεται σε κανόνες. Μπορούμε να συνεργαστούμε ε, για να δούμε πού είναι τα αμοιβαία συμφέροντα, να ενισχύσουμε τις ε, ισχύουσες συμφωνίες και να προσπαθήσουμε να βρούμε νέε συμφωνίες. Θα πρέπει όμως να σπάσουμε αυτό το φαυλοκύκλο ε, τη αντίδραση, δράση αντίδραση, α πούμε. Πρέπει να το σπάσουμε αυτό. Και ο καλύτερο τρόπο για να σπάσουμε αυτό το κακό, α πούμε, κύκλο δράση αντίδραση είναι διάλογο. Αλλά όλα εξαρτώνται από την πολιτική βούληση. Δεν είναι μαγεία ο έλεγχο των όπλων. Υπάρχουν α, συγκρούσεις στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και τις διαφορές, ουσιαστικές διαφορές επί των αρχών που υπάρχουν ε, η βασική στάση έτσι, που είναι αξιόπιστη για την αποτροπή που έχει το ΝΑΤΟ είναι πολύ σημαντική. Ε, γιατί εφόσον εμείς ξέρουμε ας που βρισκόμαστε, ξέρουν τι κάνουμε εμείς για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, οι Ρώσοι. Και εγώ που δουλεύω εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με την ε, ομάδα της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών σχέσεων με τους συναδέλφους του ΟΗΕ είναι πολύ σημαντικό για μένα. Όλοι συνεργαζόμαστε για, πάνω σε διάφορα προγράμματα που αφορούν τα μικρά όπλα. Θέλουμε να μειώσουμε την παράνομη διακίνηση όπλων ε, και τις, ε, τα πυρομαχικά τα οποία μπορούν να υπάρχουν παντού και να δημιουργούν αιστείες ανασφάλειας. Ξέρω πώς θα αποφύγουμε τον ψυχρό πόλεμο. Το έχουμε, καταφέρει τον αποφύγουμε και άλλη φορά. Ελπίζω οι πολιτικοί μας ηγέτες να έχουν την σοφία να μας απαλλάξουν από κάτι τέτοιο. Thank you, gentlemen. Σας ευχαριστούμε κύριε λέει η Πρόεδρος. Και τώρα, συνάδελφοι, θέλετε να λέτε το λόγο. Α, ο κύριος Γκάλερ. Όχι. Εκτός μικροφώνου ο κύριος Γκάλερ. Κύριε Φανόρντεν τότε. Κύριος Βανόρντεν. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω πρόεδρε τους ε, δύο προσκεκλημένους μας, τους δύο μιλητές, γιατί ήταν ακριβείς, ήταν ευσύνοπτοι, γιατί αυτό δεν το βλέπουμε κάθε μέρα να έχουμε τόσο αξιόλογες ε, εισηγήσεις στην Επιτροπή μας. Κάτι πάρα πολύ βασικό. Αν για κάποια ιστορική αναδρομή, ξέρουμε ότι πολλές φορές η αλληλεγγύη στη Δύση τρεμοσβήνει και ότι έχουν υπάρξει κάποιε ρογμέ και οπότε σε αυτήν την περίπτωση πάνε το εκμεταλλευτεί η Ρωσία. Και σήμερα στο G7 ε, δεν υπήρξε καμία ομοφωνία όσον αφορά το τι απόκριση θα δοθεί στην Ρωσία σε σχέση με τα γεγονότα της Συρίας. Υπήρξε επομένως ε, αυτό το έλλειμμα αλληλεγγύης. Άρα είναι δύσκολο το πώς θα μπορέσουμε οι δυτικές δημοκρατίες να τα βρουν όσον αφορά το ποια θέση θα υιοθετήσουν έναντι της Ρωσίας και πώς θα ε, αντιδράσουμε τον καλύτερο τρόπο. Τι λέτε. Mr. Στέτινα. Κύριε Στέτινα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας να μιλήσετε την μου γλώσσα. Συζητούμε για τα συμβατικά όπλα. Όμω, τι γίνεται στην Ουκρανία. Δεν πρόκειται για συμβατικό πόλεμο. Και ξέρω πολύ καλά τι έγινε στην ε, Μαριούπολη, στα νότια της χώρας και στο Σιρόκινο. Πολλά χρόνια. Οι Ρώσοι λέγουν το τι γίνεται εκεί στην ε, πρώτη γραμμή. Και αυτοί που τώρα πολεμούν για τη χώρα, τώρα τσακώνονται και παραπονιούνται. Και λένε ότι πολεμάνε μια ώρα, μετά σταματάει η ανταλλαγή των πυρών και μετά ξανασυνεχίζει. Έτσι κάτι τέτοια λένε. Αυτά λένε οι Ουκρανοί εκεί και λένε μα γιατί θα πρέπει να ζήσουν κατά αυτόν τον τρόπο. Πώς να μείνουν. Δεν είναι τραγικό. Γι' αυτό σας ρωτάω κύριε Μόσινκοφ. Ποιος είναι ο ρόλος του ΟΑΣΕ όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κύριε Άλμπερκ, μας μιλήσατε για την αποτροπή και τον ρόλο του ΝΑΤΟ όσον αφορά την αποτροπή. Για την Ουκρανία μπορείτε κάτι να κάνετε σχετικά. Thank you. πρόεδρος επίσης και ε, πες μας, ο κύριος Ζέμκε, σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ήταν ε, σωστή αφετηρία για μια συζήτηση. Οπότε και εγώ θα υποβάλω κάποιες ερωτήσεις. Συζητούμε για τον έλεγχο των αξιοπλισμών για τα συμβατικά όπλα. Αλλά πού είναι τα όρια μεταξύ συμβατικών και μη συμβατικών όπλων. Ποια είναι η διαχωριστική γραμμή. Εδώ έχουμε εξελίξεις που έχουν επισυμβεί. Άρα τι γίνεται. Δεύτερον. Έχουμε μια σειρά συνθήκων, συμφωνιών για την μείωση των εξοπλισμών και έχουμε διάφορους περιορισμούς που έχουν προβλεφθεί, που έχουν συμφωνηθεί και αν ρίξει κανεί μια ματιά σε αυτές τις συνθήκες και συμφωνίες, θα διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται. Δεν τηρούνται επακριβώς. Εσείς που τα υποπτεύετε όλα αυτά, για πέστε μας, πού γίνεται η πιο έντονη κούρσα εξοπλισμών από πλευράς τεχνολογικής, τι γίνεται. Γιατί αυτό θα έχει συνέπειες στο κοντινό μέλλον. Τώρα κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Για άλλο θέμα. Είμαι Πολωνός. Και φυσικό είναι να με ενδιαφέρουν όσα γίνονται από πλευράς Ρωσίας. Τα νέα τους όπλα κλπ. κλπ. Τι είναι με το βελληνικές των πυράβλων. Αυτόν που τώρα αναπτύσσει η Ρωσία. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια ποικιλία στο βελληνικές. Έχουμε και μέσω βελληνικούς πυράβλους. Τι γίνεται, τους αναπτύσσουν οι Ρώσοι τώρα Είναι θέμα πολύ σημαντικό. Θέμα ασφάλεια για την Ευρώπη και την Πολωνία. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Δυστυχώ θα πρέπει ανακατεμένα να λαμβάνετε το λόγο ανεξαρτήτω πολιτικών ομάδων. Κύριε Φοντζούλικα, συγγνώμη. Ε, θα δώσω το λόγο στην κυρία Νικολάη. Ε, θα σα δώσω μετά το λόγο, κύριε Φοντζούλικα. Τώρα η πρώτη κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα συγχαρητήρια στου προσκεκλημένου μα για τι εισηγήσει του έχω δύο ερωτήσει πρώτο για τον έλεγχο των εξοπλισμών. Σήμερα δεν υφέτεται πλέον η κλασική προσέγγιση. Τα χημικά όπλα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορα θέατρα συγκρούσεων και κυρίως στην Μέση Ανατολή έχουν γίνει τίποτα διαβήματα για να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία όσον αφορά αυτά, τα χημικά όπλα. Άλλο. Για αυτή την πρωτοβουλία. Κύριο Στάινμαγερ. Είναι ταραγμένη και από πλευρά πολιτική, αλλά και από πλευρά τη εξέλιξη του πολέμου στη Συρία. Και κατόπιν της ε, Αμερικανικής ε, επιδρομής είχαμε τις ρωσικές δηλώσεις αλλά επίσης και τον Ιρανικό παράγοντα που αναδείχθηκε. Τι γίνεται, πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος λέτε. Άλλη ερώτηση. Τι γίνεται με την αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ όσον αφορά το ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν να υπάρξει μια κοινή πολιτική ασφαλείας θεωρεί ότι σήμερα ημέρα γίνεται εμείς στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, μέσα στο ΝΑΤΟ, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είναι σωστή προσέγγιση. Ή μήπω θα πρέπει να κινηθούμε για αυτή μας την κοινή, πολιτική ασφάλεια εκτός ΝΑΤΟ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Κύριε Φουντζούλικα. Um, uh, Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι καινούργια κούρσα εξοπλισμών που γίνεται παγκοσμίω. Τρομερή ένταση. Όπω αρχέ δεκαετία του 60. Και έχουμε ακόμα προκλήσει και απειλές που έχουν κατά τη γνώμη μου πολύ κλασική μορφή. Τι προστασία έχουν τώρα οι χώρες της Δύσης έχουν το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, το ΝΑΤΟ και ιδίω το άρθρο υπαριθμών 5 τη σχετική συνθήκη. Και το έχω πει αυτό επανειλημμένα και σα το επαναλαμβάνω αξιότιμη προσκεκλημένη ότι το άρθρο 5 όμως δεν μας καλύπτει 100% όπως και θα γνωρίζετε. Προβλήπου το 5 ότι το ΝΑΤΟ πρόκειται να αναλάβει τη δράση η οποία κρυφεί ότι είναι αναγκαία, όπως θα κριθεί ότι είναι αναγκαία, ούτως ώστε να αποκαταστήσει και να διατηρήσει την ασφάλεια. Όμως, όμως, όπως ξέρετε, ε, αυτό πάνε να πει διπλωματική πίεση και φτάνει μέχρι χρήση πυρηνικών. Ε, άρα δεν ήρθε η ώρα να θωρακιστεί καλύτερα το άρθρο 5 να αναβαθμιστεί. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει εδώ πρόβλημα, υπάρχουν παραθυράκια σε αυτή τη ρύθμιση και γεωγραφικά τι πάει να πει επίθεση. Δεν έχουμε δώσει ακόμα ορισμό του τι είναι, γιατί δεν είναι μια αυθεντική πραγματική επίθεση κατά μέλους του συμφώνου. Δεν προβλέπεται ακόμα στην εργαλειοθήκη μας. Πού είναι ο ορισμός του υβριδικού πολέμου αυτόν που ειναι ο ορισμος του υβριτικου παντού η Ρωσία, προπαγάνδα, διαφθορά, επιθέσεις, τα πράσινα στρατιωτάκια οι δορυφόροι, έχει αναπτυξεί δυνάμεων στο Πακιστάν, Συρία, παντού, εφηνίδια. Α, υπήρξε κενό εξουσίας στην ε, Συρία, οπότε ευθύ αμέσω το εκμεταλλεύτηκαν. Ε, την αδράνεια τον είπα και του ΝΑΤΟ, για να τα λέμε με το όνομά τους. Εμείς είμαστε οι συμμεφορεί. θα είναι εδώ να μην μπορούμε κάτι να κάνουμε. Έχουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά πρέπει να ξέρουμε πού πάμε. Μα δεν θα πρέπει να σεβαστούν τις ε, συνθήκες οι Ρώσοι. Αυτό το πιο σημαντικό είναι η realpolitik. Εμείς πώς θα απαντήσουμε σε όλα αυτά. To my I would... Αλλά όπως και οι συνάδελφοι λέει και εγώ θέλω κάτι να σας ρωτήσω. Όσον αφορά την αποτροπή. Remarks, I would like to, to deliver first Οπότε, για πέστε μου. Ποιες είναι δεχόμενες πολιτικές συνέπειες και αποτελέσματα του διαλόγου. Γιατί το θέμα ήταν πώς θα πετύχουμε τώρα έχουμε καλύτερες συνθήκες όσον αφορά του τι θα γίνει με τους διαφωνούντες. Καλά, καλύτερα είναι τώρα από ότι επί Έχουν καλύτερη τύχη της αντιπολίτευσης. Τα είδαμε αυτά. Από πρώτο χέρι. Όμως δυσκολεύουν τώρα τα πράγματα. Α, κοιτάξτε για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Κρυμαία. Τι γίνεται με ολόκληρες ομάδες του πληθυσμού, όπως τους τάτρους της ε, Κρυμαίας. Τι γίνεται με τους της αντιπολίτευσης στην Ρωσία. Και έχουμε ένα σωρό τώρα ψηφισμάτων. Καλά δεν λέμε μόνο για, για την δολοφονία του Νέμτσοφ. Οπότε, κάπως γίνει μια στροφή στα πράγματα σήμερα. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά. Επίσης, τι κάνετε, υποπτεύετε, παρακολουθείτε τα γυμνάσια, τις σωτιές ασκήσεις των Ρώσων. Τώρα έχουν καινούργια τακτική όσον αφορά τις ασκήσεις αυτές. Μπορούμε να ασκήσουμε αποτελεσματική εποπτεία και παρακολούθηση με την ίδια σειρά. Πάρετε το λόγο κύριε. Κύριο Φροντζούρικα κάτι λέει εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Βεβαίω κάποιε από αυτέ αφορούσαν ξεκάθαρα τον ΝΑΤΟ, οπότε δεν θα τι απαντήσω. Πρώτα απ' όλα έχουμε την δήλωση του κυρίου Φανόρντεν για την δυτική αλληλεγγύη και το πόσο εξασθενεί. Προφανώς ο ΣΑ έχει 57 κράτη που συμμετέχουν και παρά το ότι υπάρχει συντονισμός στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει πάντα μια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να προσθέσω ε, ισχυρή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει έλλειψη αλληλεγγύης όταν μιλάμε για τον έλεγχο όπλων και την τρέχουσα κατάσταση ε, ασφαλείας. Και θα έλεγα ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια η κρίση της Ουκρανίας έχει επηρεάσει πολύ τις ε, συζητήσεις, αλλά δεν θα έλεγα ότι η έλλειψη αλληλεγγύης φαίνεται κάπου σε μας. Οπότε ανεξαρτήτως του πώς έχουν οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες και με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης στην Βιέννη, με όλα τα κράτη-μέλη, υπάρχει θα έλεγα μια πολύ ισχυρή θέση η οποία αρθρώνεται κάθε εβδομάδα και πάλι μεμονωμένα κράτη υπάρχουν γύρω από το τραπέζι, οπότε υπάρχει περιθώριο συζητήσεων, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά απόψεων όταν μιλάμε για την ασφάλεια της Ευρώπης. Οπότε για το πρώτο αυτό θέμα θα έλεγα ότι ε, εμείς στην Βιέννη τα βλέπουμε κάπως διαφορετικά από ότι εσείς ε, στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Στέτινα για το θέμα που θέσατε της, των αποστολών παρακολούθησης ε, στην Ουκρανία. Α, δεν είναι τώρα η θέση μου εμένα να μιλήσω για αυτό. Εγώ ήρθα εδώ για να μιλήσω για τον έλεγχο συμβατικών όπλων. Οπότε δεν θα μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά θα πω το εξή ότι η ειδική αποστολή παρακολούθησης λειτουργεί εκεί και πάλι με βάση μια συνενετική εντολή 57 κρατών. Και η εντολή που έχουν έχει σαφώς ε, διαμορφωθεί για να έχει μόνο έναν ρόλο παρατήρησης και πηγαίνει μόνο μέχρι εκεί που θέλουν να το αφήσουν τα κράτη. Οπότε ε, κάθε μέρα είναι στην γραμμή αντιπαράταξης και διαβάζουμε τις εκθέσεις τους ε, και κάθε μέρα είναι πιο κοντά στο να κινδυνεύσουν και χαιρόμαστε που δεν έχουν πάθει τίποτα αλλά είναι 1.400 άτομα, που δεν είναι πολλά βεβαίω, θα σκεφτούμε παραδείγματο χάρη μια ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ που θα είχε χιλιάδε ανθρώπου. Ε, εντάξει, έχει και διαφορετικό ρόλο βεβαίω. Αλλά δεν έχει επιτραπεί κάτι τέτοιο εκεί. Οπότε αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή ο είναι το μάξιμο που μπορεί να γίνει και συζητάμε το πώς μπορεί να προχωρήσει, αλλά προφανώς ε, και διάφοροι παίκτες επιτόπου αποφασίζουν τι περιθώριο έχει ο ΑΣΕ. Κύριε Ζέμκε, ρωτήσατε για τα όρια του συμβατικού και μη συμβατικού ελεγχού, το όπλο, συμβατικών και μη όπλων. Είναι σαφές, νομίζω, το τι ορίζουν οι συνθήκες, γιατί εκεί πέρα ορίζονται και τα οπλικά συστήματα. Εάν τα κράτη θέλουν να πάνε παραπέρα, από τα τωρινά όπλα και υπάρχει μια όθηση για κάτι τέτοιο γιατί υπάρχει τεχνολογική πρόοδος στο κυβερνοδιάστημα ή μη επανδρομένα αεροσκάφη που θα μπορούσαν να προσθεθούν στην εξίσωση αυτή αλλά δεν υπάρχει ακόμα πλήρης συμφωνία των 57 κρατών όπως είπε και ο Βίλιαμ κάθε βήμα βασίζεται στην αμοιβαιότητα. Οπότε δεν είναι το τι θέλουμε εμείς να κερδίσουμε, αλλά και ταυτόχρονα να παραχωρήσουμε. Και εκεί όπου υπάρχει μια ανισορροπία στις δυνατότητες ή στην τεχνολογική πρόοδο ε, που υπάρχει, ε, δεν είναι κανείς διατεθειμένος βεβαίω να αποκαλύψει τα μυστικά του στην άλλη πλευρά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στοιχείο αυτό των διαπραγματεύσεων. Και προφανώς δεν έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ για να έχουμε πιο ποιοτικά στοιχεία εκεί πέρα. Και για την κατάσταση Θα το απαντήσει και αυτό ο συνάδελφος για την κατάσταση στην Πολωνία, για τα μέσου βεληνικούς ε, βλήματα με πυρηνικές δυνατότητες. Θα το απαντήσει και αυτό ο συνάδελφος. Κύριε Νικολάη, ρωτήσατε για τα χημικά. Ο ΑΣΕ επειδή εστιάσατε στη Μέση Ανατολή, κοιτάξτε, εμείς από της αρχής έχουμε τα 57 κράτη. Δεν είναι κάποιο από αυτά στη Μέση Ανατολή και στη Μεσόγειο. Συνεργαζόμαστε με κάποια από αυτά, αλλά έχουμε και ένα πρόγραμμα και εντολή να εργαστούμε επί της απόφασης 15-14 του Συμβουλίου Ασφαλείας του όπου βοηθάμε τα κράτη που συμμετέχουν και κάνουμε πολλή δουλειά, πραγματικά χάρη στην Κεντρική Ασία και στα Βαλκάνια, για να φτιάξουν τα εθνικά σχέδια δράσης ε, και να εργαστούν προς την εφαρμογή τους. Και αυτό βεβαίως περιλαμβάνει και τα χημικά. Βιολογικά, ε, χημικά και πυρηνικά όπλα. Ε, τα στηρίζουμε αυτά, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ανάλογα προγράμματα, π.χ. στην Ουκρανία και όλοι συμμορφώνονται με τη Σύμβαση Περιχημικών όπλων. Όλοι είναι συμβαλόμενα μέρη. Οπότε κατά από αυτή την ομπρέλα των χημικών προσπαθούμε να λειτουργήσουν τα πράγματα πρακτικά. Για την πρωτοβουλία του κυρίου Στάνμαϊρ. Ε, λέτε ότι είμαστε σε καιρούς ε, δύσκολους. Εγώ θα έλεγα ότι οι καιροί ήταν ήδη τέτοιοι, γι' αυτό προέκυψε η πρωτοβουλία Στανμάιερ. Ήδη στον έλεγχο των όπλων ήταν δύσκολη κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια αρκεί μια ιστορική αναδρομή και θεωρώ πως η τρέχουσα κρίση απλά επιδίνωσε τις ε, αντιφάσεις και τις αντιρρήσεις κάποιων κρατών, αλλά δεν θα συμφωνούσα ότι ξαφνικά τώρα επιδεινώθηκε η κατάσταση σε σχέση με ένα χρόνο πριν ειδικά εάν δούμε τον έλεγχο Οπότε προσπαθούμε να βρούμε μία διέξοδο και πάλι την Παρασκευή που μας πέρασε ήταν όλα τα κράτη που συμμετέχουν στον διάλογο ε, διατεθειμένα να ανοίξουν τα χαρτιά τους για να επιτύχουμε μία συμφωνία. Για το ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ, αυτές οι ερωτήσεις με αφορούν. Ε, μία ερώτηση της κυρίας Πρόεδρου για τις ασκήσεις ad hoc. Πολύ σημαντική γιατί είναι μία διάταξη στο έγγραφο της Βιέννης, ε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ότι εάν δεν προειδοποιεί κανείς τα στρατεύματά του εκ των προτέρων και θέλει να κάνει μια άσκηση ετοιμότητας, υπάρχει μία, άσκηση, μία διάταξη που λέει ότι ε, δεν χρειάζεται να να ειδοποιηθούν οι άλλες χώρες 42 ε, μέρες πριν, αν είναι μια άσκηση που αφορά πάνω από 9.000 ε, στρατιώτες ε, και άρματα κλπ. Αυτό το ήθελαν και οι δυτικοί τότε, έτσι, το 1990, γιατί δεν θέλαμε να ενημερώνουμε όλες τις άλλες χώρες, αλλά τώρα είμαστε κάπως πιο ευαίσθητοι, καθώς ειδικά η Ρωσία κάνει αυτές τις ξαφνικές ασκήσεις, και είναι βεβαίως ανησυχητικό, αλλά δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη να πούμε «Α, τώρα να βγει η διάταξη γιατί δεν μας βολεύει». Και γεγονό είναι ότι τότε αφορούσε βεβαίως αμυντικές ασκήσεις, ασκήσεις ε, για την πυραυλική άμυνα κτλ. Αλλά για αυτές τις περιπτώσεις είχε γραφτεί. Οπότε τώρα η κατάσταση είναι διαφορετική, θέλουμε να αλλάξει και βεβαίως η Ρωσία οπωσδήποτε θα μας πει ότι αυτό στρέφεται εναντίον μας, εάν ε, αφαιρεθεί αυτή η διάταξη. Οπότε είναι οπωσδήποτε ένα στοιχείο που μας ανησυχεί και υπάρχει κάποια δυσπιστία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιλύσουμε. δεν υπάρχει συνένεση ε, π.χ. για να υπάρχουν μεγαλύτερες ποσοστώσεις, δηλαδή να γίνουν ξαφνικές ασκήσεις, αλλά ειδοποιήστε μας και καλέστε μας. Ε, είναι με επιλογή, αλλά δεν συμφωνούν τα 5-7 κράτη. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ για τις θαυμάσιες ερωτήσεις. Χαίρομαι που μου τις κάνετε. Τεσσερά μισή ή πέντε χρόνια πριν, όταν ξεκίνησα να δουλεύω στο ΝΑΤΟ, δεν φανταζόμουν ότι θα υπάρχουν τέτοιε ερωτήσει. Τώρα όλο και περισσότερο ενδιαφέρονται για τέτοια θέματα. Χαίρομαι για αυτό το επίπεδο λοιπόν ενδιαφέροντο και συμμετοχή. Για το πρώτο ερώτημα για την αλληλεγγύη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν πηγαίνω στη Βιέννη και ακούω τις ε, δηλώσεις ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά για την Ουκρανία. Είναι θαυμάσιες, είναι δυνατές, είναι ομόφωνες, μια φωνή και κάθε φορά βάζουν τους Ρώσους στη γωνία. κάθε μέρα <laughs> πάντως πρέπει να τσεκάρουμε σε τι φάση είναι οι Αμερικανοί, μήπως έχουν έτοιμοι να εκστρατεύσουν αντίον του διαστήματος του το G7, το G7 δεν είναι τόσο ενοποιημένο όσο ήταν. Κοιτάω τι γίνεται και στο ΝΑΤΟ, όπω εξετάζω τι γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπω μια μεγάλη αποφασιστικότητα. Θα ήθελα να συνεχίσουμε έτσι και να την ενισχύσουμε μάλιστα. Εγώ όμως στο ΝΑΤΟ αισθάνομαι ότι η συνένεση είναι μεγάλη μας δύναμη και όπως είπα και στη Βιέννη η ομοφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα της Ουκρανίας είναι εντυπωσιακή. Χαίρομαι για αυτές τις δηλώσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διατλαντική συνένεση ήταν η πιο σημαντική πράξη. Ε, όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά για το αδιέρετο της ασφάλειας, κατάλαβα ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να λυθούν τα προβλήματα της ε, Ευρώπης χωρίς τη συμμετοχή της Αμερικής και του Καναδά. Και αυτή η διατλαντική συνένεση είναι πολύ σημαντική. Το ΝΑΤΟ το επιθυμίζει συνάχη συνέχεια. Και ελπίζουμε αυτό να ξαναεμφανιστεί στην διάσκεψη του ΝΑΤΟ, να ξαναεπαναδιατυπωθεί. Για τη δήλωσή σας, Η δουλειά που κάνει η ειδική αποστολή ε, της Ουκρανίας είναι πολύ σημαντική και θα ήθελα η συμφωνία κατά ψωπυρός να παρακολουθείται πιο σοβαρά ε, και να υπάρχουν και ασφαλιστικές που το ώστε να μην ξανααρχίσουν οι εχθροπραξίες, γιατί βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις ε, συμβαίνει συνέχεια. Επίσης, ε, το... Ε, υπάρχουν συστήματα, ηλεκτρονικά συστήματα για να ελέγχουν τους εξοπλισμούς η αποτροπή τώρα μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας για την Ουκρανία καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε διαφορετικούς πλανήτες. Οι χώρες που θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ ε, πριν γίνουν πλήρη μέλη ε, εκτίθενται, αντιμετωπίζουν πολλά ρίσκα. Ε, έχουμε πολλές περιπτώσεις υβριδικών πολέμων που προωθούνται, διαβάζουμε σε εφημερίδες, ε, διαβάσαμε τι έγινε στο Μαυροβούνιο. Είναι μια τρομερή κατάσταση αυτή των υβριδικών πολέμων. Ε, μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα για την Ουκρανία, αλλά μια και δεν είναι μέλο του ΝΑΤΟ, πάντα υπάρχουν όρια στο τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, Όπω ε, είχαμε και περιορισμού στο τι μπορούσαμε να κάνουμε στι ε, διάφορε σειράξει ανά την Ευρώπη τα τελευταία 15-20 χρόνια. Η επόμενη ερώτηση. Ε, υπάρχουν τα συμβατικά όπλα και τα πυρηνικά όπλα. Ποια είναι η διαφορετική γραμμή και ποια είναι η τομή και η ένωση. Ε, η γραμμή μεταξύ του συμβατικού πολέμου και του πυρηνικού πολέμου. Μπαίνουμε για πρώτη φορά σε μια περίοδο που για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες ακούμε ε, να εκτοξεύονται πυρηνικές απειλές στα πλαίσια συμβατικών πολέμων. Ε, διάφοροι απειλούν θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα. Η όλη έννοια, όλη η ιδέα ας πούμε, της αποκλιμακοποίησης ε, από τη χρήση των πυρηνικών έχει υποσκάπτονται. Επίσης, η Ξέρουμε ότι η Ρωσία μπορεί να απειλήσει την Ευρώπη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, λένε μην ανακατευτείτε. Ε, το έλεγαν μάλλον παλιά. Ε, γιατί τότε θα σας επιτεθούμε. Γι' αυτό θέλαμε να ξεφορτωθούμε αυτά τα, αυτούς τους πυράβλους μεσαίου βεληνικούς. Και τη στιγμή που μπούσαμε να του ανοιχνεύσουμε ήταν στο τσακ για να ε, χτυπήσουν τι ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε. Ήταν αποσταθεροποιητική η κατάσταση. Ελπίζω να μην ξαναμπούμε σε αυτή τη φάση που είχαμε επί εποχή Σοβιετική Ένωση. Αλλά αυτή ο διαχωρισμό ανάμεσα στα συμβατικά και στα πυρηνικά όπλα θα πρέπει να θα τον ξαναδούμε. Ε, εμείς το, οι Ρώσοι το είχαν ξεχάσει. Εμεί δεν το είχαμε σκεφτεί για πολλά χρόνια. Όπω επίσης και το θέμα του ελέγχου των εξοπλισμών. Εμείς στο ΝΑΤΟ δημιουργήσαμε μια επιτροπή για να εξετάζει τα πυρηνικά όπλα και το πρώτο πρόβλημα που θέλαμε να λύσουμε είναι ε, τα, τους πυράβλους μεσαίου βεληνικούς. Εν συνεχεία τα τακτικά όπλα και μετά το 1987 και μέχρι το 1990 το ΝΑΤΟ σκέφτηκε τη συνθήκη που θα απόκλει όλα τα τακτικά όπλα, όλα τα στρατηγικά όπλα θα σταματούσαν να υπάρχουν όλοι οι πύραυλοι μεσαίου βελληνικούς θα ε, ρυθμίζονταν από τη συνθήκη INF και μετά θα μπαίναμε στα τακτικά όπλα. Ο Μπούς και ο Γκορμπατσόφ τελικά συμφώνησαν να μην αντιμετωπίσουν τα τακτικά όπλα στα πλαίσια μιας συνθήκης. Αλλά τώρα, εάν θα κάνουμε διάλογο με τη Ρωσία, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την απειλή από τα τακτικά όπλα. Ε, ελπίζω να τα αντιμετωπίσουμε αν ποτέ αποφασίσει διάλογο σοβαρό η Ρωσία μαζί μας για το, τη μείωση των εξοπλισμών. Πού είναι ε, ως η σημαντικότερη κούρση εξοπλισμών. Είναι στον Κάφκασο. Ε, Αζερβαϊτζάν ε, μπορεί να αποσταθεροποιηθεί η συνολικότερη περιοχή Ιράν, να μπει και η Τουρκία μέσα. Γι' αυτό δεν εγκαταλείπουμε τη συνθήκη CFE. Ξέρουμε ότι δεν την έχουν τηρήσει στον Κάφκασο, ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα συμμόρφωσης, αλλά καλύτερα να υπάρχει ένα νομικά δεσμευτικό, μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δράσουμε παρά να μην έχουμε τίποτα. Για την INF θα πρέπει να ξαναρυθμίσουμε αυτό το θέμα. Ε, παραβιάζει η Ρωσία τη συνθήκη αυτή. Ε, είναι άμεση απειλή για την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων. Ε, και θα πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία ελέγχου των ε, εξοπλισμών η Ρωσία. Είναι ε, προϋπόθεση. Θα πρέπει να τηρήσουν όλες τις ε, διεθνείς συμφωνίες τους. Ε, όμως η απροθυμία τους να συζητήσουν το θέμα αυτό με τις ΗΠΑ είναι άσχημη εξέλιξη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Νικολάη, κύριε Νικολάη, χημικά όπλα. Η, Ρωσία ως εγκύτρια της ασφάλειας της, της Ρωσίας δεν έκανε θαυμάσια δουλειά, έτσι ε, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τα, τις αποθήκες όπλων κτλ. Τι έγινε τελικά. Ξέρουμε ότι οι στρατιωτικοί της ε, Συρίας ε, ρίχνουν χημικά όπλα σε αμάχους. Ε, θα έπρεπε να υπάρχει καταγραφή και από τους Ρώσους και να κατακρίνουν τους Σύριους ότι δεν έχουν σεβαστεί τις διεθνείς δεσμεύσεις τους. Ε, θα έπρεπε να καταστρέψουν τα, τις αποθήκες πυρομαχικών και τα συστήματα ε, εξαπόλυσης όπλων κτλ. Επίσης, ε, κύριε Ρόμπιν, χρειάζεται διάλογο όταν ε, υπάρχει πρόβλημα. ε, όταν σταμάτησαν την επικοινωνία σοβιετική και Αμερικανοί ε, με, για οποιοδήποτε θέμα, ας πούμε, εναρίας κυκλοφορίας, ε, για να μην υπάρξει σύγκρουση μεταξύ να μην χτυπήσουν ένα στον τον Αυτό, αυτό με ανησύχησε εμένα. Όσο περισσότερο διάλογο έχουμε, τόσο καλύτερα. Και ειδικά όταν υπάρχουν ζωφερές ε, και προβληματικές περιοχές, χρειάζεται αυτό. Τώρα, ΝΑΤΟ ή Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ σας δίνει το πλαίσιο, της, ε, την κατάρτιση, τις ιδέες, δεν σας δίνει όμως ε, στρατιωτικές δυνάμεις. Αν θέλετε στην Ευρώπη στρατιωτικές δυνάμεις, εντάξει. Χρησιμοποιήστε αυτά που κάνει καλά ο, ε, το ΝΑΤΟ, δηλαδή έχετε τη δομή, την, ε, το διοικητικό μηχανισμό, ας πούμε, το, την κατάρτιση και είμαστε πολύ αξιόπιστοι στο να παράγουμε σενάρια. Ο, θα μπορούσε να συμφωνήσει, πούμε, η Ευρώπη Επίσης θέλω να έχει πιο έντονη ασφάλεια η Ευρώπη, αλλά θέλω να χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες δομές του ΝΑΤΟ παρά να παράγει τις δικές της δομές και να υπάρχουν επικαλύψεις. Αν μια χώρα θέλει να ενταχθεί και να πει ότι είναι θέμα του άρθρου 5, έχουμε προβλήματα στο, με το άρθρο 5. Για το, έχουμε το άρθρο 3 που λέει ότι θα πρέπει όμως και εσείς να μπορείτε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Το άρθρο 4 είναι αυτό που λέει ότι ο τύπος σας ανησυχεί, έλατε στο άρθρο να το πείτε. Για το άρθρο 5, το αν μια χώρα αποφασίζει ότι είναι υποαπειλή, ε, τότε θα πρέπει να συζητήσουμε το άρθρο 51 της χάρτας του ΟΗΕ. Αυτό δεν σημαίνει μαζική επίθεση με συμβατικά όπλα, μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα, ακόμα και βιβλικό πόλεμο. Ένας, ένας από τους λόγους που ε, χρησιμοποιούμε τον όρο υβριδικός πόλεμος είναι ότι Ξέραμε επί ψυχρού πολέμου τι συνέβαινε, τι συνέβαινε τότε με την προπαγάνδα, με όλα τα άλλα ε, παραφερνάλια, ας πούμε. Ε, δεν θέλουμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, ας πούμε, γι' αυτό χρησιμοποιούμε τον όρο υβριδικός πόλεμος. Επίσης, δεν θέλω να είναι πολύ λεπτομέρειε το άρθρο 5, γιατί μειώνεται η ελευθερία των χωρών του ΝΑΤΟ. Cyber, you know what cyber, uh, cyber is another area where... Κυβερνοχώρους. Ορισμένοι το θέτουν ως νέο θέμα. Ε, παλιά το λέγαμε σαμποτάζ. Υπήρχε από παλιά. Και αν συνδέεται μια κυβέρνηση, τότε ε, η κυβέρνηση, αν προκαλεί το σαμποτάζ ή την τρομοκρατία, έχουμε τα ίδια προβλήματα με την δεκαετία του 80. Ε, δεν μπορούσαμε τότε να επιθετεθούμε στη Σοβιετική Ένωση. Το θέμα είναι ότι ως κοινωνίες αποφασίσαμε να ξεχάσουμε να εξασφαλιστούμε, ας πούμε. Και ποια είναι η... το σημείο ευαλωτότητάς μας, ας πούμε, είναι αυτό. Ε, εάν μέσω του σαμποτάζ αυτού, ας πούμε, σε αυτά τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά συστήματα, ας πούμε, μπορεί να πλήξει τους πολίτες του κτλ. Ε, αν αποσταθεροποιεί την ε, κοινωνία σου, δεν χρειαζόμαστε νέε έννοιε. εντάξει. Αυτό υπάρχει εδώ και αιώνες αυτή η απειλή. Τέλος, Πρόεδρε. Η τελική πράξη του Ελσίνκη. Η ανθρώπινη διάσταση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ. Ε, τι γίνεται ε, με τους ε, διαφωνούντες, οι οποίοι βοήθησαν στο να πέσει το σοβιετικό καθεστώς. Ο, είναι ένα μάθημα που διδάχτηκε πολύ καλά, έμαθε πολύ καλά ο Πούτιν. Και η δημοκρατία, η, η καταπολέμηση της διαφθοράς, οι ελεύθερες εκλογές και τα λοιπά, όλα αυτά απειλούν τη δική του θεώρηση των πραγμάτων για τη Ρωσία. Ο ρόλος της ΟΑΣΕ είναι να εξασφαλίσει την ελευθεροτυπία, τις ανοιχτές εκλογές λοιπά, την ε, δημοκρατία και τα λοιπά. Και ελπίζουμε να επηρεάσει και την ε, Ρωσία ε, και την κεντρική Ασία. Υπάρχει και μια τελική διαφάνεια, ε, θα ήθελα να την αναρτήσετε, που δείχνει τις ασκήσεις από το 2009 έως το 2016. Εγώ παρακολουθώ τις ε, στρατιωτικές ασκήσεις στην Ατλαντική περιοχή γενικά. Και χαίρομαι που το έγγραφο της να υπάρχει, που υπάρχει ο, η ΟΑΣΕ, ο, η γιατί έχουμε πληροφορίες. Επίσης, χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ αυτές τις ασκήσεις για να εντοπίσει τα προβλήματα και έχουμε κανόνες για να λέμε εκ των προτέρων ότι ε, ας πούμε μην ξεχνάτε την ε, εισβολή στην Ουγγαρία το 1956 το, και τα λοιπά ε, τις ε, απειλές στην Πολωνία το 80 και 81 που προηγήθηκαν από μαζικές, μαζικά στρατιωτικά γυμνάσιμα της, ε, στρατιω... της Ρωσίας, της Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή, το να κάνεις τέτοιες μαζικές ασκήσεις και να χρησιμοποιείς ε, τις εξαιρέσεις που υπάρχουν και να μην πεις στους άλλους τι θα κάνεις είναι πρόβλημα. Γιατί οι άλλοι μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι προετοιμασία για πόλεμο. Ε, αν κάνεις κάτι και οι άλλοι ανησυχούν και, μας λένε, και σου λένε ε, πες μας κάτι για αυτή, αλλά αυτοί που την κάνουν σου λένε Α, μια χαρά είναι όλα, δεν θα σου πω τίποτα. Υπάρχει αυτό το παραθυράκι, θα το χρησιμοποιήσω κτλ. Για να μην σου πω τίποτα, αυτό είναι ένα πολιτικό μήνυμα. Ε, γι' αυτό χαίρομαι ε, με τον ΝΑΤΟ που όταν μα ρωτάει, α πούμε, η Ρωσία, Μα τι κάνετε εσεί, ε?» και εμεί του λέμε, Κοιτάξτε, να. Ε, έχετε παρατηρητέ, ε, ελάτε ρωτήστε μα. Όταν όμω η άλλη πλευρά δεν κάνει και αυτή το ίδιο, κάτι, κάτι άσχημο συμβαίνει. Ένας, ε, σκοπός, του ελέγχου των εξοπλισμών δεν είναι να συμμορφώνονται μονίμως η άλλη πλευρά. Το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε, ας πούμε, και πότε δεν συμμορφώνονται. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώ πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε ας προσπαθήσουμε να ανακεφαλαιώσουμε όσον αφορά αυτό το σημείο. Δεν έχουμε δεύτερο ε, γύρο ερώτα απαντήσεων. Οπότε, απομένει μόνο να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη σύντομη Ενημέρωση και την ε, ζωηρή συζήτηση που ακολούθησε. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθώ σε κάτι από αυτά τα οποία είπατε για το στοιχείο εκδημοκρατισμού. Αυτό είναι αναγκαίο στοιχείο για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνη. Ακόμα και αν ο Πούτιν θεωρεί ότι είναι μια κακή ιδέα όσον αφορά το μέλλον της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εμείς το θεωρούμε ένα προαπαιτούμενο, πολύ σημαντικό, οποιοδήποτε διάλογο με τη Ρωσία. Και πάλι σας ευχαριστούμε, οπότε προχωράμε στο επόμενο σημείο ευθύς αμέσως. Colleagues, next point. Πρόεδρος. Το επόμενο σημείο σήμερα στη διάταξη, συνάδελφοι, είναι η πρώτη συζήτηση του σχεδίου γνωμοδότησης όσον αφορά τη στρατηγική της Ευρώπης για το διάστημα. Η κυρίως αρμόδια επιτροπή είναι η Ήτρε και ο σύντακτης είναι ο κύριος Τζέφρι Βανόρντεν. There are shadow rapporteurs. Οι τους και Η Γκουε, από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει ορίσει και Οπότε παρακαλούμε και την Γκουε να ορίσει και Έχετε το λόγο, κύριε Βανόρντεν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πολύ σημαντικό το θέμα θα θυμάστε ότι έχουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής του 16 για την στρατηγική του διαστήματος και ευτυχώς η Επιτροπή Βιομηχανίας αποφάσισε να συντάξει αυτή την έκθεση για το σημαντικό θέμα. Εμείς βέβαια θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής focus on. I mean, first of all, I've drawn attention to the uh, significance. Γιατί πρόκειται περί πολύ σημαντικής στρατηγικής που αφορά το διάστημα, αφορά τι διαστημικέ τεχνολογίε, τεχνολογίες, οπότε αυτό που θέλω να σας πω συγκεκριμένα αφορά τα αδύνατα σημεία, το ευάλωτον, γιατί συνεχίζονται οι προσπάθειες ε, έρευνα σε διάφορες χώρε, ιδίω σε εχθρικές χώρες, όσον αφορά κάποια συστήματα επιθετικού χαρακτήρα με στόχο κρίσιμες υποδομές, τηλεπικοινωνίες, αλλά και τα συστήματα που έχουν σχέση με τη διαστημική τεχνολογία. Άρα ε, θα πρέπει εδώ πέρα τώρα να προσέξουν, προσέξουμε περισσότερο και με καινούριο τρόπο όλα αυτά τα αναδείξουμε. Επίσης προσπαθήσαμε να τονίσουμε το πόσο χρειάζεται να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και των τρίτων χωρών και οργανισμών. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο βέβαια δεν είναι μια εντιστενή ενία υπηρεσία παρά το ότι εκεί πέρα συμμετέχουν τα τα μελη και παρά το ότι ο προπολογισμό προέρχεται κατά ένα 20% από τον κοινωτικό προπολογισμό. Τα υπόλοιπα τη προεκοδότη προέρχονται από τα κράτη-μέλη Οπότε νομίζω ότι είναι σωστό το μοντέλο της δομής και τη δίνει στην υπηρεσία διαστήματος ευελιξία και υπάρχει και ευκαιρία ευρύτερη συνεργασία με άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, όπως η Ινδία και άλλες χώρες ενδεχομένω. Έχουν διαπιστώσει προτάσει στα πλαίσια του ΟΗΕ για κάποιο είδου κώδικα διοντολογία για αυτέ τι ε, δραστηριότητε στο διάστημα. Οπότε θα πρέπει να καταλήξουν σε κάποιον τέτοιο κώδικα διοντολογίας από όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και έχουμε τώρα φτάσει στις περίπου 70 χώρες που έχουν δορυφόρους και νέα χώρες έχουν δυνατότητα εκτόξευσης σε τροχιακή θέση. Να, σε αυτά τα σημεία στάθηκα στο κείμενό μου, όπως γνωρίζετε είναι ευσύνοπτο το κείμενο και βάζω εδώ τελεία και ακούω τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε κύριε Βανόρντεν. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο κύριος Γκάλερ έχει αναλάβει να εκπροσωπήσει την κυρία Σντρογεύσκη για το θέμα Γκάλερ. Όχι, δεν μπόρεσε να έρθει ο συνάδελφος Σντρογεύσκη, οπότε ε, θα σας πω εγώ τι έχει να δηλώσει η στρατηγική για το διάστημα της ε, Ευρώπης ήταν κάτι που το περνούμε εδώ και πολύ καιρό, ιδίως έχοντας ε, υπόψη το ότι όλο ένα και περισσότερο εμπλέκεται σε δραστηριότητες τέτοιες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τη στρατηγική 14 ε, με 2020, οπότε επενδύσαμε 12 δις όσον αφορά τα προγράμματα Galileo και Copernicus και είχαμε περίπου 30 εκτοξεύσεις ε, που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη 20 Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί ένας από τους πιο σημαντικούς αποδέκτες ε, των προϊόντων της σχετικής βιομηχανία στην Ευρώπη. Αυτή η στρατηγική ε, προβλέπεται σε αυτό το σύντομο κείμενο για το τι συγκεκριμένε δράσει θα ληφθούν τα επόμενα χρόνια και έχουμε τώρα την γνωμοδότηση του κ. Φανόρντεν που είναι σωστή αφετηρία για συζήτηση. Όμω θα πρέπει να επιφέρουμε κάποιε αλλαγέ. Θα πρέπει να δούμε αυτή τη στρατηγική από πλευράς εξωτερικής δράσης της ε, Ένωσης και από πλευράς ασφαλείας. Μ' αρέσει ότι υπάρχει εδώ αυτή η παράγραφος για την ασφάλεια των διεθνικών συστημάτων καθευτών, αλλά και όσον αφορά την υποδομή που οδηγεί σε αυτές τις δραστηριότητες. Επίσης, ε, συμφωνώ με αυτή την ε, μνήμα της προσπάθειας καταδίκης των επιθετικών όπλων αλλά επίσης και την προσπάθεια της κατάρτισης κώδικα διοντολογίας στα πλαίσια του ΟΗΕ. Αυτό το οποίο λείπει από το κείμενο είναι δεν αναφέρεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική διαστήματος εννοείται ότι είναι αρμοδιότητα εθνική. Όμως η συνθήκη της Λισαβόνας ξεκάθαρα ορίζει ότι μπορεί να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δικές της δραστηριότητες αυτό κάνει και με επιτυχία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, προτείνω να βάλουμε και μία παράγραφο που να αναφέρεται στι δυνατότητε του Γαλιλαίου και ιδίω του Κοπέρνικου όσον αφορά την ασφάλεια μέσω παρατηρήσεων δεδομένων, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η εξωτερική δράση της Ένωσης, ιδίω στα πλαίσια της ΚΕΠΑ. Πώς και πω και ανυπόμονα περιμένω τη συνεργασία με τον κύριο Βανόρντεν. Αυτά μου είπε να σα διαβάσω, λέει ο κύριος Γκάλερ. Πρόεδρο. ευχαριστούμε κύριε Γκάλερ. Ο κύριος Φρουντζούλικα θέλει να λάβει το λόγο. Είστε και εσεί και ο δισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Βανόρντεν για το σχέδιο κειμένου. Έχουμε εδώ πολλές προσεγγίσεις του εισηγητή με τις οποίες συμφωνούμε ιδίω για το ότι έχουμε αυξανόμενη σημασία του διαστήματος και των τεχνολογιών ιδίω αφορά πληροφορίες, επιτήρηση, αναγνώριση κλπ. Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε το πόσο ευάλωτες είναι αυτές οι, τεχνολογίες. Ευάλωτες από επιθέσεις κρατικές και μη κρατικές. Άρα εδώ πρέπει υπάρχει θέμα ασφάλειας είναι πολύ βασική διαστημική τεχνολογία για την ασφαλεία μας αλλά και την οικονομία μας και γι' αυτό. Άρα είναι σημαντικό να προαγάγουμε μια τέτοια αυτονομία στις υπηρεσίες που αναπτύσσουμε για το διάστημα. Τα τονίζει αυτά ο κ. Βανόρντεν ότι έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλούς ε, εμπλεκομένους πολλούς παράγοντες οι οποίοι έχουν πολλές δυνατότητες αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος από τα προγραμματά τους τα διαστημικά. Άρα θα πρέπει να βρεθούν κάποιοι κοινοί κανόνες για να είναι το διάστημα να είναι προσβάσιμο σε όλου και ασφαλές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν προτείνει να υπάρξει κάποιος ε, κώδικα διοντολογία για αυτές τις δραστηριότητες, όπως λέει και ο εισήγητης, να ενθαρρύνουμε τις προσπάθειες του ΟΗΕ, να υπάρξει συμφωνία για αυτό το θέμα και να υπάρξει και κάποιο ε, κώδικας με εκούσια προσχώρηση, συνεργασία χρειάζεται στη διεθνή σκηνή για αυτά και να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μα με τον ΝΑΤΟ, με τι ΗΠΑ και άλλε χώρε ούτω ώστε τα θέματα ασφάλειας και άμυνας να προσεχθούν. Επίσης θα πρέπει να προσπαθήσουμε και μέσα στην, Ευρωπαϊκή, στην Ευρώπη στρατηγικό, πολιτικό ε, συμφέρον, αναβαθμίζουν δυνατότητες, βιομηχανικά, τεχνολογικά, γιατί η στρατηγική αυτονομία θα ωφελήσει όχι μόνο τους συμπολίτες και τα μέλη αλλά και τους εταίρους. Αν έχουμε όλο το φάσμα των στρατηγικών δυνατοτήτων, έτσι θα γίνουμε ισχυρός εταίρος και του ΝΑΤΟ, σίγουρα. Επίσης, να υπάρξει νοτόζα του ΝΑΤΟ να μπορεί να έχει δυνατότητες ε, εκτόξευσης συστημάτων. Πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό, το, ώστε να έχουμε και συνέργειες, να βοηθεί και η απασχόληση σε σχέση και με άλλες ε, κρατικές πολιτικές. Τα κράτη-μέλη μέσω της Επιτροπής ε, της Υπηρεσίας Διευθύματος θα πρέπει να προχωρήσουν προς αυτό το μέτωπο. Μπράβο και ας συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, λέει στον εισηγητή ο κύριος Φροντζούλικα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τώρα η κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτό το σύντομο κείμενο του Τζέφρι είναι σημαντικό το θέμα. Δεν έχω όλη την έκθεση, έχω μόνο την γνωμοδότηση στα χέρια μου. Πάντως, θα ήθελα να προσθέσω ένα-δύο σημεία όσον αφορά την στρατηγική διαστήματος πρώτα-πρώτα. Πόσο σημαντική είναι η χρήση του διαστήματος όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας όσον αφορά την επιτήρηση, την εποπτεία, την παρακολούθηση. Έτσι μπορούμε να έχουμε σαφείς πληροφορίες και έτσι να έχουμε καλύτερη λήψη αποφάσεων. Επίσης, να έχουμε το σύστημα διπλής χρήσης. Σημαντικό. Να αντιμετωπίσουμε το hacking και πρέπει αυτό να θεωρηθεί εκείνο που θα αντιμετωπιστεί. Αλλά βέβαια έχει οικονομική σημασία να δυνατοτήτων των ε, στρατηγικής διαστήματος και πρέπει να υπάρξουν εξελίξεις που θα είναι οικονομικά αποδοτικές. Σημαντικό αυτό. Και επίσης τελευταίο αλλά σημαντικό, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη-μέλη πρέπει να αναπτύξουν μια πραγματική συνεργασία αλλά και σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών για να αποφύγουμε επικαλύψεις αλλά και κούρσα εξοπλισμών στο διάστημα. Μπορεί να κατεβάσουμε κάποιε τροπολογίε, αλλά εν γέννη συμφωνούμε με το κείμενο του κ. Βανόρδεν. Ευχαριστούμε κύριε Νικολάη, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα, κ. Σίντρεκ. Ο κ. Τάραντ. Ίντρεκ Τάραντ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Πρώτα πρώτα ευχαριστούμε και τον κύριο Βανόρντεν για αυτή τη γνωμοδότηση. Μπέρα την πολιτική διαστημάτωση επιτροπής. Πρώτα πρώτα κάτι το οποίο στην Εστονία ήταν κλασική σκέψη όταν ήμουν νέο, το 62. Λέγανε, τότε ακούσατε, βγήκανε οι Ρώσοι στο διάστημα και η απάντηση ήταν «Ε, τι, όλοι τους. Ναι, βλέπετε, στην Εστονία πάντα είχαμε στρατηγική για το διάστημα. Αλλά τέλος πάντων, όσον αφορά την ευρωπαϊκή στρατηγική, οι πράσινοι γενικώ συμφωνούμε. για τα σχετικά με την πολιτική διαστήματος. Πάντως εργάζομαι και στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών, οπότε και θεωρώ υποχρεωσή μου να σας υπενθυμίσω ότι μιλούμε για κάποια δις ευρώ. Άρα θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να δούμε κατά πόσον αυτές οι επενδύσεις αποδίδουν. Αν μέχρι το 2020 επενδύσουμε 12 δις, να προσέξουμε πολύ στο τι απόδειξη θα έχουν όλα αυτά τα χρήματα. πλευρά πρασίνων θα έπρεπε να δούμε το κατά πόσον μπορούμε για το διάστημα να διαθέσουμε τον προϋπολογισμό, την του Twitter. Βέβαια, ε, αυτές οι προσπάθειες που συζητούμε έχουν σχέση και με την ασφάλεια και την άμυνα και εμείς είμαστε υπέρ. Πάντως υπάρχει μια κάποια σύγχυση. Κατά πόσο δηλαδή μπορούμε κάτι να κάνουμε μέσω διαστήματος για τον έλεγχο των συνόρων και την μετανάστευση. Η καλά, η μετανάστευση βέβαια γίνεται στη γη, όχι στο διάστημα. Να, γιατί χρειάζονται πράσινες πολιτικές. Άρα πολύ ωραία όλα. Και αναφέρει την ε, πρωτοβουλία κ. Βανόρδεν όσον αφορά τον, τη διεθνή προσπάθεια κάποιου κώδικα διοντολογίας για τις διαστημικές δραστηριότητες. Και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό δεν το ανέλαβε ως προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και καλύτερα τώρα το Κοινοβούλιο να διορθώσει τα κακοσκήμενα στη δουλειά της Κομισιόν. Τώρα φτάνουμε στο διατάφτα σε αυτό το αξιολογικό κείμενο, Βαν Όρντεν έχει ε, πει για τις κυβερνοεπιθέσεις εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε τίποτα στο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις αλλά επίσης και το άλλο το την ε, σκέψη για, τις, για τους ελέγχους των εξαγωγών και ξαναγυρίζουμε στο στο αστείο αυτό για το ότι γινόταν το 62. Ευχαριστώ. Κύριος Νάρτ. Ευχαριστώ. Ε, συμφωνα, συμφωνώ γενικά με την πρόταση του κυρίου Βανόρντεν, που είναι και σύντροφος, αλλά πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση δεν είναι απλή. Έτσι, στο σημείο 3 Μιλάμε για την ε, απειλή, για το πρόβλημα που θέτουν οι χώρες όπως η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν και για τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγονται για τις δικές μας υποδομές και επικοινωνίες. Αυτό είναι συνέπεια ανάμεσα στη σύγκρουση μεταξύ της ΗΠΑ και της Ρωσίας. Οι ΗΠΑ έχουν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα, το να ισχυριστούμε ότι η Ρωσία και αφήστε την Βόρεια Κορέα που είναι εγκληματικό κράτος εξορισμού ότι έχει τελείως διαφορετικό πρόγραμμα από το πρόγραμμα που έχει ε, μία από τις δύο μεγάλες δυνάμεις, όπως και η Κίνα το έχει ας πούμε, είναι σαν να υπάρχει το δικαίωμα του να επιτίθεσαι και να καταστρέφεις τις επικοινωνίες. Ε, και αυτό το δικαίωμα το έχουν μόνο οι φίλοι μας. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα όμως. Γι' αυτό λοιπόν το σημείο 3 είναι συνέπεια ανάμεσα στην αντίφαση, ανάμεσα σε δύο δυνάμεις που κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Το να θεωρήσουμε ότι είναι ο διάβολος η Ρωσία ε, λόγω αυτών που κάνει, τη στιγμή που κάνουν ακριβώς τα ίδια οι Αμερικάνοι, δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα. Ε, γιατί ούτω ή άλλω δεν υπάρχει και συγκεκριμένη αναφορά και στην Κίνα. Εκτό και αν θεωρήσουμε ότι η Κίνα είναι σύμμαχο, που δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Δεύτερο σημείο, προβληματικό σημείο 4. Το να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την εκτόξευση δορυφόρων ε, από τους Ρώσους, δεν νομίζω ότι μας οδηγεί σε λάθος κατεύθυνση. Ε, από τη μία ε, θέλουμε μια στρατηγική συνεργασία που επηρεάζει την ασφάλειά μας. και έτσι απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο από κοινέ αξίες. Η Ρωσία βασικά απομακρύνεται. Αυτό σημαίνει ότι κόβουμε όλες τις γέφυρες, ακόμα και τις τεχνολογικά δυνατές. Ε, σε αυτή την περίπτωση την εκτόξευση δορυφόρων από τους Ρώσους, όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και με την Αριάδνη, ας πούμε, που είναι ευρωπαϊκός, ευρωπαϊκή βάση ας πούμε, για την πυράβλων, που έχει πολλά λάθη, πολλά προβλήματα. Δεν νομίζω ότι ότι με αυτόν τον τρόπο ε, θα αντιμετωπίσουμε τις διαφορές μας με τη Ρωσία. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κόβουμε όλες τις γέφυρες, ε, θα φτάσουμε σε ένα καταπληκτικό ψυχρό πόλεμο, όπου δεν θα υπάρχει τίποτα από άλλο κατηγορίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είναι λάθος κατεύθυνση αυτή. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς απέναντι στους Ρώσους, αλλά ούτε πρέπει να επανέλθουμε στον ψυχρό πόλεμο. Ε, σαν να είμαστε σε φάσεις στον προθάλαμο του πολέμου του ψυχρού πολέμου φαντάζομαι. Ε, αυτά για τα σημεία 3 και 4. Για τα σημεία 3 και 4 έχω πρόβλημα. Με τα υπόλοιπα όμως συμφωνώ απόλυτα. Ευχαριστώ. Πρέπει να κλείσουμε το σημείο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα ζητήσω από τον κύριο Φανόρντεν ε, να σχολιάσει αυτές τις παρατηρήσεις που άκουσα. Και να απαντήσει και όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα προσεκτικά του σχόλια. Πολλά, πολλά από αυτά ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Ε, το μόνο που θέλω να πω είναι το εξή. Ορισμένοι μίλησαν για τα οικονομικά ωφέλη του διαστήματο. Φυσικά, τα γνωρίζω. Αλλά σε αυτή τη γνωμοδότηση μην ξεχνάτε ότι είναι μια γνωμοδότηση που εξετάζει πολύ στενά τα θέματα άμυνα και ασφάλεια. Δεν εξετάζει τι οικονομικέ πτυχέ. Ε, το Ήτρε ασχολείται με αυτά, η Επιτροπή Ήτρε. Ε, κατά τα άλλα, σας ευχαριστώ για τα σχόλια και τη συνεργασία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι ο Απρίλιος στις 24 Μαρτίου μέχρι τις 6... Απρίλιο, συγγνώμη, μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες φυσικά. Σας ευχαριστώ για αυτό το σημείο. Παρακαλώ, μείνετε για το επόμενο σημείο. Πρέπει να περιμένουμε μια στιγμή, λίγα λεπτά, γιατί οι επόμενοι ομιλητές μας, ο Διευθυντής Κένεθ Ντίν, είναι στο δρόμο και έρχεται. Colleagues, please be seated. Okay. It is my pleasure. Καθίστε. Με χαρά καλωσορίζω έναν ε, γνωστό μας ε, στην Επιτροπή, τον κύριο Δίν, ε, Διευθυντή της μη στρατιωτικής δυνατότητας προγραμματισμού στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και ο στόχος μας ε, σήμερα λοιπόν είναι η πλατφόρμα στήριξης αποστολής για ένα πρώτο βήμα προς ένα διακλαδικό κέντρο ερωτηματικό. Επίση ο κύριος Ντίν θα είναι εδώ πέρα και αύριο στην συνεδρίασή μας. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Έχουμε καθυστερήσει λίγο λόγω τεχνικών προβλημάτων. Χωρίς άλλη χρονοτριβή, λοιπόν, να δώσω τον λόγο στον κύριο Ντίν. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για τα καλά σας λόγια. Πάντα χαίρομαι που έρχομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως υπάλληλος βεβαίως θέλω μια κατεύθυνση από εσάς για το τι κάνουμε στην ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Λοιπόν, θα ήθελα να φερθώ, όπως είπε η κυρία Πρόεδρε, στην πλατφόρμα στήριξης ε, των αποστολών και αν δούμε τον τίτλο, βλέπουμε πως πρόκειται για μια διαδρομή. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να αναφέρω μια διαδρομή, γιατί η διαδρομή είναι από το που βρισκόμαστε αυτή την στιγμή, στο που θέλουμε να πάμε, δηλαδή σε ένα διακλαδικό κέντρο να ξεκινήσω λοιπόν από το τέλος της διαδρομής, εάν μου επιτρέπετε, το τι σημαίνει δηλαδή ένα διακλαδικό κέντρο. Ένα διακλαδικό κέντρο θα μας δώσει μια ελάχιστη γνώση και τεχνογνωσία που θα είναι διαθέσιμη για κάθε μη ε, στρατιωτική αποστολή σε τρεις υπήρους όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή θα δημιουργούσε ε, έναν ευέλικτο πάροχο υπηρεσιών που θα επιτρέψει την βέλτιστη χρήση των πόρων κατά την κατάρτιση των αποστολών. Επίσης ε, θα επιταχύνει τις ε, διαδικασίες πρόσληψης ε, προσωπικού. Και θα ενισχύσει οπωσδήποτε την ορθή διαχείριση και την χρηστή διαχείριση και την εμπειρία εξπόστ βεβαίω για το πώς θα σεβόμαστε τον δημοσιονομικό κανονισμό και τη γενική αρχή της ορθής ε, δημοσιονομικής διαχείρισης και θα μας επιτρέψει να έχουμε ακόμα περισσότερα συμβόλαια πλαίσιο με τρόπο συνεπή για να ανταποκριθούμε σε όλες τις απαιτήσει μη στρατιωτικών αποστολών θα αποτελέσει ένα κέντρο επιμελητίας ε, και θα εναρμονίσει τις διαδικασίες για την στήριξη των αποστολών Εν ολίγης λοιπόν ένα τέτοιο κέντρο είναι κάτι το θετικό και βεβαίως είχαμε και την έκθεση του Συμβούλου πριν από λίγα χρόνια που ενθάρρυνε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε όμως φτάσει εκεί, αυτό είναι το τέλος της διαδρομής, οπότε να κάνω λίγο προς τα πίσω. Ε, αυτή τη στιγμή είμαστε στην αρχή. Ποια είναι λοιπόν η ζήτηση. Το Νοέμβριο του 2016 είχαμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Παγκόσμια Στρατηγική για την εφαρμογή της ε, ΚΕΠΑ και εκεί πέρα λέει επιλέξει. Ζητάει από την υπηρεσία εξωτερική δράση να ενισχύσει τις ε, πτυχές εκείνες οι οποίες είναι κοινέ για όλες τις αποστολές, να υπάρξει μια πλατφόρμα ως ε, μέρος προσπάθειας να αναπτυχθεί ένα κοινό διακλαδικό κέντρο. Οπότε τα κράτη-μέλη ακόμα αναμένουν από εμένα και τους συναδέλφους στην υπηρεσία εξωτερικών να προωθήσουμε το θέμα. Τι είναι λοιπόν η πλατφόρμα. Θα είμαι ειλικρινής. Είναι ένα πολύ μικρό πρώτο βήμα προς την διαδρομή ενός διακλαδικού κέντρου. Είναι μικρό από, σκοπιά, από άποψη μεγέθους Αυτή τη στιγμή ε, έχει δύο μονάδες, μία στην δική μου διεύθυνση που αποτελείται από 7 άτομα στην ε, μη στρατιωτική δυνατότητα σχεδιασμού και βεβαίως υπάρχουν και ε, άλλοι 8 συνάδελφοι στην Κομισιόν. Πρόκειται λοιπόν για έναν πολύ περιορισμένο αριθμό καθώς αρχικά είχαμε ζητήσει 27 άτομα για ένα μικρό τέτοιο κέντρο και 48 άτομα για ένα πιο μεγάλο κέντρο, οπότε μιλάμε για ελάχιστο αριθμό, οπότε έχουμε το 25% του διακλαδικού αυτού κέντρου και ανάλογα πρέπει να κινηθούν και οι προσδοκίες μας. Αλλά ξεκίνησε η ε, πλατφόρμα με την απόφαση του Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2016. Οι 7 συνάδελφοι λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουν, είναι τέσσερις ειδικοί πληροφορικής, δύο ειδικοί επιμελητίας και ένας ανθρωπίνων πόρων. Να σας πω τι κάνω λοιπόν αυτή τη στιγμή. Σας είχα πει λοιπόν πως α, τελικός μας στόχος είναι ένα πλήρες κέντρο. Ε, οι συνάδελφοι λοιπόν αυτή τη στιγμή δημιουργούν ε, τους εξυπηρετητές ε, και ένα μια διαδικτυακή πύλη προσπαθούν να δημιουργήσουν διαδικασίες ε, πληροφορικής ε, και καλύτερη επικοινωνία και συστήματα διαχείρισης εξοπλισμού. Επιπλέον εξετάζουν τις διάφορες εφαρμογές ε, πληροφορικής. Έχουμε εννέα αποστολές αυτή τη στιγμή που κάνουν εννέα ξεχωριστά πράγματα και δεν είναι αποδεκτό αυτό την σήμερον ημέρα. Πρέπει να εργαστούμε πολύ πιο έξυπνα και αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ, ήδη εδώ, Δηλαδή, εγώ αν είχα έναν ειδικό σε μία αποστολή, ε, θα μπορούσα να περιμένω να πάει σε μία άλλη αποστολή και να ξέρει το τι θα αντιμετωπίσει από πλευράς διαδικασιών, πρωτοκόλων Οπότε χρειάζεται κάπου να υπάρχει αυτή η πείρα σε ένα σημείο κεντρικό για να ενισχύουμε αυτούς τους συναδέλφους για να ξέρουν πώς θα κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα. Γιατί οι επιχειρησιακές, επιχειρησιακά αποτελέσματα κάθε αποστολής είναι τόσο καλά όσο η στήριξη αυτής της αποστολής. τότε θέλω οι συνάδελφοι να είναι έτοιμοι όπου πηγαίνουν, να πηγαίνουν σε μια αποστολή οργανωμένη. Και δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα. Δεν έχω στόχο να ασκήσω κριτική στις τρέχουσες αποστολές. Λοιπόν, όσον αφορά ακριβώς ε, την πλατφόρμα υπάρχουν και οι δύο συνάδελφοι που ασχολούνται με την επιμελητία και αναπτύσσουν αυτή τη στιγμή κάποιου όρου αναφοράς ε, και συζητούν με την Κομισιόν το τι μορφή θα πρέπει να έχει. Ίσως θυμάστε πως είχαμε πει πως ε, ότι ακριβώς ε, θέλαμε να έχουμε μια αποθήκη αν θέλετε όπου θα αποθηκεύουμε τον εξοπλισμό, π.χ. τα οχήματα Λοιπόν, οι συνάδελφοι δουλεύουν με βάση την απόφαση του Συμβουλίου. Τρεις χώρες ζήτησαν αυτή την αποθήκη. Η Σουηδία επέτυχε και ακριβώς κάνουμε μια αξιολόγηση με βάση τον σχετικό πυλώνα για να δούμε ότι υπάρχουν όλες οι οικονομικές δομές πριν δώσουμε λεφτά. Και αυτό λοιπόν είναι εξελίξη. Και υπάρχει κάποιος ο οποίος αναπτύσσει ένα σύστημα ανθρωπίνων πόρων όπου βεβαίω αν θεωρούμε ότι οι άνθρωποι είναι ο σημαντικότερος πόρο χωρί τι κατάλληλε πληροφορίε και ένα σύστημα πληροφορική και μια κατάλληλη πολιτική ανθρωπίνων πόρων, δεν θα έχουμε το κατάλληλο άτομο στο κατάλληλο μέρο, στην κατάλληλη στιγμή και θα είναι λιγότερο αποτελεσματικέ οι αποστολέ μα. Και τέλο. Θέλουμε ακριβώ να καθοδηγήσουμε και τι ε, πρωτεύουσε ε, έτσι ώστε να μπορούν να βρίσκουν του κατάλληλου ανθρώπου νωρί. Και αυτή είναι δική μα υποχρέωση. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε καλύτερε διαδικασίε, ε, περιγραφέ του αντικειμένου, να ξέρουν το τι περιμένουν τα κρατημέλη, γιατί του τελευταίου 12 μήνε καταφέραμε να ελεγχιστοποιήσουμε τις περιγραφές αντικειμένου από χίλιες ε, κάτω από 197 γιατί νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι πάνε σε αποστολές κάνουν λίγο πολύ τα ίδια πράγματα δηλαδή το κράτος δικαίου είναι κράτος δικαίου εντάξει υπάρχουν διαφορετικές προκλήσεις αλλά στη σκοπιά της στήριξης παραδείγματο χάρη είναι οι αρμόδιοι για τις προμήθειε είναι αρμόδιοι για τις προμήθειε παντού όπως και οι αρμόδιοι για το κράτος δικαίου και άλλες ειδικότητε και νομίζουμε πως μια πλατφόρμα θα μπορούσε να μας βοηθήσει περαιτέρω στην εξέλιξη μιας ομοιοτυπίας ε, στις αποστολές. Οπότε, όπως είπα, 7 συνάδελφοι, 4 πληροφορικάροι, 2 ε, στην επιμελητία, ένας ε, στους ανθρώπινους πόρους Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά να κάνουμε και όσον αφορά τις δικές μας δεξιότητες αλλά και τους πόρους που θα χρειαστούν αλλά όπως ξέρετε τα διαφορετικά θεσμικά όργανα έχουν διαφορετικές απόψεις για το διακλαδικό αυτό κέντρο. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ και είμαι στην διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις, σχόλια κτλ. Σας ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Τώρα θα δώσω τον λόγο στους συναδέλφους. Πρώτος ο κύριος Γκάλερ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τις δηλώσεις σας. Άκουσα από διάφερους συναδέλφους που είχαν πάει στις αποστολές το πόσο δύσκολο είναι να έχουν τα διάφορα πράγματα που χρειάζονται εκεί και πόση ώρα χρειάζεται. Οπότε μου φαίνεται ότι είναι λογικό να κάνουμε αυτό το οποίο προτείνετε, αλλά και τον τελικό σας στόχο βεβαίως. Κάντε το λοιπόν και προσπαθήστε και πείτε μας ε, ή πείτε σε μένα ποιοι είναι αυτοί που σας ε, φέρνουν προσκόμματα. Και αν είναι στη δικιά μου τη χώρα θα έρθω σε επαφή μαζί τους. Είναι κάτι το λογικό αυτό το οποίο ζητάτε, κάνει καλύτερα την δουλειά, εξοικονομεί κόστος και θα πρέπει να το στηρίξουμε. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν έχει γίνει τόσο καιρό. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Van Orden. Κύριος Van Orden. Thank you very much, Madam Chairman. Um... Πάντοτε ευπρόσδεκτος εδώ ο κύριος Ντίν. Στη Ραμάλα τα είπαμε τελευταία φορά. Κάπου εκεί τέλο πάντων. Έχω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα. Μας είπατε ότι χρειάζεστε να υπάρξει συνέχεια, να υπάρξει πυρογνωμοσύνη. Άρα πού το πάτε. Να υπάρχει κάποιο είδους τέτοια προσπάθεια που να αναπτύσσεται να είναι δυνατόν να αναπτυχθεί όποτε χρειάζεται φιλόδοξη η ιδέα. Επίσης, τι λέτε για την αποτελεσματικότητα των αποστολών. Επενδύουμε πολύ χρήμα στις αποστολές αυτές. Και πολλές φορές η αποστολή ξεκινάει και μετά την ξεχνάμε. Ωραίες οι παρουσιάσεις PowerPoints, αλλά μετά λέμε πού το το αποτέλεσμα το χειροπιαστό. Άρα μπας και θα πρέπει να έχουμε κάποιους μηχανισμούς ώστε να ε, αντλούμε συμπεράσματα από το παρελθόν, μαθήματα και να αποτελεσματικές ο αποστολές. Κύριε Ντίν, λέει Θα μπορούσατε τώρα να απαντήσετε και μετά να έχουμε άλλο κύριο να το απαντήσουμε. Πρώτα πρώτα για τον κύριο Γκάλερ. Ε, έχει άλλε. απόψεις, έχει αλλάξει άποψη τώρα, τέλο πάντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορώ βέβαια εγώ να μιλήσω αντί των κρατών μελών, αλλά τέλος πάντων αλλά για την ΚΕΠΑ δεν έχουμε ε, κάποια νέα εντολή. Επομένως, τι να πω. Αλλά οπωσδήποτε και χρειάζεται αυτό το κέντρο σχεδιασμού των επιχειρήσεων. Έτσι είναι. Είναι ωφέλιμο. και οικονομικά. Βεβαίω και υπάρχουν επικρίσεις. Και ακριβώ αυτό θα θεράπευε την έλλειψη ευελιξίας που υπάρχει. Ε, ευχαριστώ για καλά σας λόγια κύριε Βανόρντεν. Ναι, ναι, στην Ραμάρα τα είχαμε πει τότε υπό την προηγούμενη μου αρμοδιότητα. Δεν θα το ήθελα αυτό, εδώ ήταν το ιδιώδες για οποιονδήποτε επικεφαλής αποστολής ή οργανισμού. Ακριβώς χρειάζεται βοήθεια από όλες τις απόψεις σε μια αποστολή. Αυτό θα ωφελούσε αυτό το κέντρο σχεδιασμού και υποστήριξης. Άρα, από τη μια μεριά έχουμε το επιχειρησιακό κομμάτι, από την άλλη μεριά το οργανωτικό. Σε κάθε περίπτωση. Επομένως, το ιδιώδες ποιο είναι. Παρά τις επικρίσεις για τις ε, μη στρατιωτικές αποστολές, το να μην έχουμε ταχεία ανάπτυξη. Να έχουμε όμως σωστή απόκριση. μπορούμε να αναπτυχθούμε όπου χρειάζεται. Και έτσι θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες που υπάρχουν. Το θέμα είναι βέβαια τι θέλει και πόσο γρήγορα θέλει να αναπτυχθούν τις δυνάμεις η χώρα που γίνονται αυτά. Ε, βέβαια το θέμα είναι με τι μηχανισμό θα γίνει αυτό. Να, αυτά θα κάνει αυτό το κέντρο σχεδιασμού. Αλλά αυτό θα είναι δυνατόν μόνο εάν είναι διαθέσιμο το προσωπικό. Να υπάρχει ετοιμότητα. Μόνο έτσι. Και αυτό που είπατε κύριε Βάνορδεν. δεν έχουν πάντα τους ιδιώδεις που είναι έτοιμοι να αναπτυχθούν. Δεν λέω ότι έχουμε τους χειρότερους, αλλά αν δεν υπάρχει ετοιμότητα, πώς να έχουμε ταχύ ανάπτυξη. Να μια λύση. Να είμαστε έτοιμοι να υπάρχει η δυνατότητα με το CPCC να υπάρχει και τον προτέρων συμφωνία του σχετικού κράτους και κάποιος που διατίθεται που είναι να πηγαίνει όπου χρειάζεται. Έτσι μπορεί να γίνει η ανάπτυξη γρήγορα. Να υπάρχει κάποιο είδου διαρκής δυνατότητα. Το θέμα δεν είναι πόσοι θα είναι αυτοί. Ας είναι 15-16. Ας μην είναι παραπάνω. Να υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, ούτως ώστε αυτή λίγη αλλά σημαντική, με την επιμελητία, την ασφάλεια κλπ. να είναι έτοιμοι να πάνε. Πέραν του κανονισμού των δημοσιονομικών. Άρα θα πρέπει να κινηθούμε με ευφία. Οπότε να δούμε το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκό στρατός ή σε δεύτερη φάση οι εξειδικευμένε ε, ομάδες και έτσι να ενισχύουμε αυτούς που θα αναπτυχθούν εκεί καταρχήν ταχύς ανάπτυξη και κατόπιν ενισχύσεις με φυσιολογικές διαδικασίες ε, ανάθεσης. Άρα υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα πάγιας, διαρκούς φύσεως. Και έχετε δίκιο για την ε, αποτελεσματικότητα. Αν είχαμε εδώ τους επικεφαλείς, θα σας λέγανε πόσο τους παρενοχλώ, πόσο τους κολλάω. Αυτό τους λέω ότι θα πρέπει συνεχώς να πετύχουν κάτι, να πετύχουν κάτι χειροπιαστό. Δεν είναι μόνο το πολιτικό θέμα. Να έχουν κάποιο είδου σχέδια εφαρμογής να αφορούν τα άτομα αλλά και τις ομάδες αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια. Και κάθε μήνα να μου αναφέρουν τι πάει στραβά και τι πάει καλά. Και τους λέω να είναι ειλικρινείς, να μου λένε τι δεν πάει καλά. Έτσι μόνο θα έχουμε την ε, πολιτική υποστήριξη από τις Βρυξέλλες. Οπότε αυτό κάνουμε κύριε Βαν Όρντεν. Είναι υπόλογες οι αποστολές και εγώ επίσης αυτό κάνω με τις εντολές για τις αποστολές που δίνω. Να πιάνουν τόπο οι επενδύσεις που κάνουμε σε αποστολές. Να, Στόχο μου λοιπόν είναι ότι θα πάνε όλα καλά και, και με την Επιτροπή σα εδώ στο Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστούμε, Διευθυντή, κύριε Διευθυντά. Οι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν και άλλε παρεμβάσεις. Όχι. Πολύ ωραία. Θα θέλα να... Να κλείσουμε αυτό το θέμα της σημασία διάταξης. Κύριε Ντίν, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Φαντάζομαι ότι θα έρθετε και αύριο. Το επόμενο σημείο στην μέση διάταξη γίνεται κυκλισμένο των θυρών. Θα ήθελα οι να ελέγξουν ότι μόνο τα άτομα που πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα παραμένουν.